Παρακαλώ, χρόνο φίδου. Ναι. Προφανώς θέλει να απαντήσει ο κύριος Άγνιου. Ήταν ξεκάθαρα τα δεδομένα ότι ο αέρας μετέφερε τον ιό όπου φυσούσε και έτσι κατέστησε ακόμα και πιο δύσκολη την ε, αντιμετώπιση της επιζωοτίας και εσείς που προέρχεστε για το North Northumberland ε, που έχει καταγραφεί ότι πρέπει η ταφή να γίνεται μέσα σε 24 ώρες δεν αρκεί η αποτέφρωση το πρόβλημα ήταν ότι έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο η συγκέντρωση στους χώρους αποτέφρωσης των ε, ε, σφαγίων των ζώων, των πτωμάτων των ζώων και γι' αυτό υπήρχε, υπήρξε ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος. Ο Λόρδος λοιπόν ε, έπρεπε να έχει εισακουστεί. Βεβαίω και εν τέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε το σφάλμα τη, επιτρέποντας τη ταφή σε συγκεκριμένου όμως χώρου, όχι μέσα στην ίδια την εκμετάλλευση, πολλές φορές μέχρι και 300 χιλιόμετρα μακριά, δηλαδή έπρεπε τα πτώματα των ζώων να μεταφέρονται σε φορτηγά, πολλές φορές υγρά ε, πτωματικής προελεύσεως ε, κυλούσαν στο δρόμο γιατί ξεχύλιζαν από τα φορτηγά ήταν η κατάσταση απαράδεκτη και αφόρητη. Παρακαλώ, πολύ σύντομα, ναι, και θέλετε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, Κύριε Μπράνον. Ναι, προφανώς και ήταν αφόρητο. Εσείς όμως ισχυριστήκατε ότι η αποτέφρωση διέδωσε την επιζώτια. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη προς την κατεύθυνση αυτή και θα ήθελα να μου παρουσιάσετε τέτοιου είδους αποδείξεις. Ότι η αποτέφρωση προξένησε διάδοση της επιζωτίας. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπράμαν. Σίγουρα μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα και έχουμε και τους ειδικού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαντάζομαι θα συγκεντρώνουν και εκείνες τις πληροφορίες, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να επεκταθούμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Καλύτερα να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Το 6 αναβάλλεται και λίγο αργότερα, μέχρι όταν έρθει η κυρία Μακαντάιρ. Και πάμε στο σημείο 7, τη νέα συμμαχία για την επιστημιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Ανάπτυξης. Η συντάκτρια γνωμοδότης Επιτροπής Γεωργίας είναι η κυρία Μόλι Σκοτ Κάτο. Αλλά ούτε και η κυρία Σκοτ Κάτο έχει έρθει. Μήπως θα μπορούσαμε να διεκπαιρεώσουμε το σημείο 8, το θέμα του κυρίου Αντριέ, αν είναι παρόν ο κύριος Αντριέ και αν δεν έχει πρόβλημα. Ωραία. Θα περάσουμε στο 8 θα ακούσουμε την παρουσίαση του Αντιπροέδρου μας, του κυρίου Αντριέ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι και παρόν και πανέτοιμος να μας ενημερώσει για το πολύ αυτό σημαντικό το θέμα, πώς μπορεί η κοινή γεωργική πολιτική να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ήπεθρο και στην ανάπτυξη της Ήπεθρου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της ανάπτυξης της Ήπεθρου Η βρίσκεται στην καρδιά τη Ευρώπη. Ε, καλύτερα όμω το θέμα θα μα το παρουσιάσει ο αρμόδιο ε, συντάκτη τη γραμματότητα, ο κύριο Αντρία. Παρακαλώ, κύριε Αντρία. σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντω, ε, προέβλεπα να κάνω κάποιε μικροδιευθετήσει στην παρουσίασή μου αυτή, ενώ θα είχαν πάρει το λόγο οι συνάδελφοι για τα προηγούμενα σημεία. Πάντω δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο σε καμία περίπτωση να καθυστερήσουμε περισσότερο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σα πω ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη κάπω έκθεση, γιατί ουσιαστικά έχει να κάνει με κάποιε βασικέ επιλογέ που πρέπει να κάνουμε στα πλαίσια τη κοινή γεωργική πολιτική. Ξέρετε ότι συνήθω προσεγγίζουμε την κοινή γεωργική πολιτική και την απασχόληση με πολλού διαφορετικού τρόπου από πολλέ διαφορετικέ σκοπιέ. Όσον αφορά τώρα την υφιστάμενη γεωργική κατάσταση, και λαμβάνοντας υπόψη επίσης και όλες αυτές τις κρίσεις οι οποίες πολλαπλασιάζονται και διαρκούν πάρα πολύ καιρό και το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που εγκαταλείπουν την Ήπεθρο, θεώρησα λοιπόν λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη ότι θα πρέπει αυτή τη φορά να προσεγγίσουμε την κοινή γεωργική πολιτική με έναν τρόπο διαφορετικό. Δηλαδή να καταφέρουμε να μπούμε στην ουσία του ζητήματος και να απομακρυνθούμε από μια καθαρά πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσεγγίζω την κοινή γεωρική πολιτική από τη σκοπιά της απασχόλησης και θα ήθελα επ' αυτού να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και εκφράζω σαστικά την επιθυμία στο έγγραφο αυτό να μπορέσετε η μεν και η δε να θέσετε κάπως στο πλαίσιο μιας μελλοντική έκθεσης της Επιτροπής μας και ξέρω ότι μπορώ να βασίζομαι σε αυτές τις διαφορετικές οπτικές γωνίες προκειμένου να έχουμε μια σφαιρική έκθεση στο μέλλον. Αν εξετάσουμε λοιπόν την κοινή γεωργική πολιτική μέσα από το πρίσμα της απασχόλησης, ουσιαστικά καλούμεθα να αναρωτηθούμε πόσο αποτελεσματική είναι τελικά η δημόσια αυτή πολιτική, η οποία θεσπίστηκε πριν από 54 ολόκληρα χρόνια. Μια πολιτική η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 40% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια πολιτική η οποία ουσιαστικά θα έπρεπε να αντιστοιχεί σε μία από τις 10 προτεραιότητες του Πρόεδρου Γιούγκερ που είναι η απασχόληση. Παρ' όλα αυτά όμως ουδέποτε έγινε μια αξιολόγηση της κοινή γεωρικής πολιτικής, μια σοβαρή επιστημονική αξιολόγηση υπό το πρίσμα της απασχόλησης, της δυνατότητάς της δηλαδή να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Το ζήτημα λοιπόν της ε, νομιμότητας τελικά της κοινή γεωρικής πολιτικής σε σχέση με τον αντίκτυπο που έχει και στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται ή πρό, πρόκειται να τεθεί, αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά και γι' αυτό ακριβώς το λόγο νομίζω ότι δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε πλέον. Όντως, θεωρώ και εγώ ότι η κοινή γεωρική πολιτική σαφώς είναι αναγκαία, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον να παρακάμψουμε το ζήτημα αυτό το οποίο έθεσα πριν από λίγο. Ναι, μια κοινή γεωργική πολιτική, αλλά για ποια ακριβώ γεωργία. Η κοινή γεωργική πολιτική δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να περιορίζεται μόνο στην ε, κατανομή κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων στα κράτη-μέλη. Ο νόμος της αγοράς πλέον επιβάλλει πολλές φορές το να έχουμε συγκεκριμένη παραγωγή εντατική σε συγκεκριμένα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το μοντέλο αυτό έχει αποδείξει πλέον ότι δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Το μοντέλο αυτό σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε μια εδαφική εξισορρόπηση, δεν αντιμετωπίζει τα ζητήματα της δημόσιας υγείας, ούτε τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος ή τα ζητήματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Αποτελεί λοιπόν δική μας ευθύνη να επαναπροσεγγίσουμε και να θεωρήσουμε την κοινή γεωρική πολιτική βάσει συγκεκριμένων πλέον νέων στόχων. Νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την κοινή γεωρική πολιτική, αυτό το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκθέσεις μας. Το αμέσως επόμενο ερώτημα όμως πρέπει να θέσουμε είναι το πώς θα παράγουμε, πόσο θα παράγουμε και σε συνεργασία με ποιου. Πώ δηλαδή θα καταφέρουμε να πειράσουμε το ζήτημα τη απασχόληση επιτόπου. Μολονότι είχαμε πάρα πολλέ αποτυχίε στο παρελθόν και μολονότι είχαμε και τη δυνατότητα στο παρελθόν να σημειώσουμε μεγάλη πρόοδο στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Μπορούμε πραγματικά αυτή τη στιγμή να θεωρήσουμε ότι η μόνη λύση είναι η απορρίθμιση της αγοράς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο και μόνο να αντιμετωπίσουμε την κρίση την οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπω θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα άλλο μοντέλο κοινή ζωρική πολιτική. Μήπω θα πρέπει να επαναθεωρήσουμε του βασικού αυτού στόχου τη σημαντική αυτή δημόσια πολιτική που θα πρέπει να λειτουργεί υπέρ των πάντων και που θα πρέπει να προωθεί ένα νέο μοντέλο γεωργικό και κοινωνικό για το μέλλον και νομίζω ότι θα πρέπει επίση να λαμβάνει υπόψη τη τόσο την ύπεθρο, την αγροτική ανάπτυξη, καθώς επίσης και τη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Περιμένω κύριε Πρόεδρε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο προκειμένου να εμπλουτίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο το περιεχόμενο της μελλοντική αυτής έκθεσης, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί πριν το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντρία. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση της γνωμοδότησής σας. Αλλά νομίζω ότι έχετε πολύ υψηλέ προσδοκίε από την κοινή γεωρική πολιτική. Δεν μπορεί να τα ρυθμίσει όλα η κοινή γεωρική πολιτική. Πολύ συχνά λέμε ότι παρά είναι ευρεία η κοινή αγροτική πολιτική. Άλλοι δεν ασχολείται όντως με τα ουσιώδη που είναι η γεωργία, η αγορά, η κατάσταση των γεωργών στην αγορά, γιατί είναι πολλές φορές δεινή η κατάσταση των γεωργών. Και ε, επίση η γεωργία έχει επεκτάσει ε, όχι μόνο στη γεωργική πολιτική, αλλά και στην περιβαλλοντική. Εν πάση περιπτώσει, εσείς ε, το θέμα. Είναι η πρώτη συζήτηση. Ο κύριος ε, Μίγκε, κύριε Μίλερ συγγνώμη. Ευχαριστώ, θερμά πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Υποστηρίζω, δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί το θέμα της ανεργίας στην Ήπεθρο, την πρότασή της. Ωστόσο θέλω ιδιαίτερα να σημειώσω ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να προωθήσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της απασχόλησης, πράγμα το οποίο δεν πράττει. Και δεν πρόκειται εδώ για μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, όπως εσείς ισχυρίζεστε. Πρέπει λοιπόν, κατά την δική μου έποψη, να στραφούμε στα σημεία εκείνα στα οποία μπορούμε να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες που θα αντιστρέψουν τις πτωτικές ε, τάσεις της απασχόλησης στην Ήπεθρο. Προγράμματα ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Φερρυπίν, ε, το Ταμείο Ανάπτυξης της Ήπεθρου για την ανάπτυξη, απογραφειοκρατικοποίηση. Επίσης, ταυτόχρονα πρέπει να στραφούμε και προς τον νέο κτηνοτρόφο και να τον βοηθήσουμε με την απλούστευση των διαδικασιών. Οι άμεσες ε, πληρωμές για μένα δεν αμφισβούν δεν αμφισβητούνται, είναι πολύ σημαντικές για τη στήριξη του εισοδήματο και για την διατήρηση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην υπεθρό της Ευρώπης. Ε, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και γι' αυτό θα πρέπει να βελτιωθούν. Ο κύριος Χόισλινγκ παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κυρίε και κύριοι συναδελφοί. Νομίζω ότι διατυπώνονται τα σωστά ερωτήματα απόψε δεν νομίζω ότι μπορούμε ακόμα σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε να συγκεκριμενοποιούμε συγκεκριμένα ε, ζητήματα. Πρέπει να πούμε ότι όντως αμφισβητείται η νομοποίηση των άμεσων πληρωμών. να κοιτάξουμε τα επιχειρήματα και την αντιπαράθεση με τις θέσεις εργασίας που διαφυλάχθηκαν στην τελευταία περίοδο, το αποτέλεσμα, ο υπολογισμό είναι αρνητικός. Έχουμε χάσει το 50% των γαλακτοπαραγωγών στη Γερμανία, παραδείγμα, τελευταία εξαιτία. Μήπως λοιπόν πρέπει τα χρήματα να διατεθούν διαφορετικά, δηλαδή να μην είναι όλο και λιγότεροι οι γεωργοί οι οποίοι θα παίρνουν όλο και περισσότερα χρήματα. Κυρία Μίλλερ, πρέπει να τεθεί το ερώτημα. Ξεκάθαρα. Πρέπει να δούμε ίσως τα εξαγωγικές δυνατότητες, την απορρίθμιση, άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να δώσουν νέα πνοή. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε στην έκθεση του ΕΡΙΚ, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Και πρέπει στην επόμενη συνεδρίαση που θα ασχοληθεί με την ΚΑΠ να κοιτάξουμε τον τρόπο υπολογισμού αυτών των άμεσων πληρωμών γιατί δεν είναι πλέον αιτιολογημένες. Δεν είναι δυνατόν να αιτιολογούμε κάθε φορά το όλο και μικρότερο, τον όλο και μικρότερο αριθμό ε, γεωργών. Υπάρχει ζήτημα νομοποίηση, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και βεβαίω μπορούμε να συζητήσουμε ήδη στο στάδιο που βρισκόμαστε για βελτιώσει. Υπάρχει δυνατότητα για μεταφορά κονδυλίων στο δεύτερο πυλώνα για την τρέχουσα περίοδο. Αυτό θα ήταν μια ιδέα, παραδείγματι, προσυζήτησαν. Και επίση τα προγράμματα ε, ενισχύσεω θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά πόσον ε, βοηθούν, συμβάλλουν, ε, επί παραδείγματι στη δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Και βεβαίω ενδεχομένω για την προσεχή περίοδο να τα ξανακοιτάξουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει διευρυνθεί επικίνδυνο ο κατάλογος των ομιλητών, γιατί είναι σημαντικό το θέμα και ενδιαφέρον, αλλά επειδή έχουμε πάνω από 15, δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω παρά μόνο 1,5 λεπτό στον καθένα. Νομίζω ότι Άρκει πια το 1,5 λεπτό, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των ομιλητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η κυρία Ραντ Καρσία. Θα ήθελα, κύρια Άντρια, να μα εξηγήσετε τι εννοείται με αυτό το νέο κοινωνικό συμβόλαιο, γιατί αν κατάλαβα καλά αυτά που άκουσα, είναι ότι η γεωργική δραστηριότητα φαίνεται ότι περνάει με βάση την γνωμοδότησή σε δεύτερο, τρίτο πλάνο. Προτιμάται άλλα θέματα που φαίνεται ότι αντικαθιστούν τη γεωργία ως βιοποριστικό μέσο. Μιλήσατε για την ε, δέουσα χωροταξία, την ε, ιδανική χωροταξία, ε, την κοινοτική αξιοποίηση των πόρων. Μπορείτε να μας, να μας δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι εστί νέο κοινωνικό συμβόλαιο, για να καταλάβω αν θα ταχθώ υπέρ ή κατά της θέσης, γιατί απλώς διαβάζοντας το κείμενο δεν κατάλαβα καλά. Ο κύριος Νταντά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Αντριέ, διότι ξεκάθαρα στο έγγραφο αυτό παραθέτει τις ιδέες του, αλλά παρόλα αυτά έχω την εντύπωση ότι ε, διαπραγματευθήκαμε την κοινή γεωρική πολιτική το 2013, νέα διαπραγμάτευση θα γίνει το 2020 διατρέχουμε εδώ πέρα τον κίνδυνο κάθε φορά που ανοίγουμε τη συζήτηση αυτή και ενώ οι φαρμαστικοί κανόνες δεν ισχύουν για όλες τις χώρες όπως για τη Γαλλία. Πρέπει να δούμε εδώ πέρα πώς τα εφιστάμενα μέσα, τα εφιστάμενα μέσα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία. Ας μην ξεκινάμε όμως μια γενικότερη συζήτηση αυτή τη στιγμή, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί που ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήδη στα πλαίσια της δημοσιονομικής αναθεώρησης, θέλουν να αναθεωρήσουν τα κονδύλια τα οποία δίνονται στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Δεν έχουμε αρκετά κονδύλια και πολύ φοβάμαι ότι αν ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση θα μειωθούν ακόμα περισσότερα τα κονδύλια τα οποία δίνονται στην στην κοινή γεωργική πολιτική. Συγκεντρωθούμε λοιπόν πραγματικά στο βασικό ζήτημα το οποίο το βλέπουμε και στον τίτλο αφού τον γράφω εργασία. Πώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κοινή γεωργική πολιτική για να ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων απασχόληση σε αγροτικέ περιοχέ. Α συγκεντρωθούμε σε αυτό. Κυρία Σλάιρ. Yeah, Als u kijkt naar dit onderwerp, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστήσω τον κύριο Αντριέ. Το 2020 πραγματικά να ρωτιούνται οι αγρότες το τι θα γίνει, αν τελικά θα πρέπει να επανδιαπραγματευτούμε εντελώ την κοινή γεωργική πολιτική. Α μην ξεχνάμε ότι ένα από του στόχου τη κοινή γεωργική πολιτική είναι και η ασφάλεια, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και εκτό. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η απαραίτητη χρηματοδότηση θα δίδεται στους γεωργούς, προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν να επιτελούν την εργασία τους. Το 2020 σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δούμε ούτε απαλωτριώσεις ούτε μείωση των κονδυλίων και δεν νομίζω ότι δημιουργούνται και τόσες πολλές θέσεις απασχόλησης από την κοινή γεωργική πολιτική. Πόσες θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν όχι μόνο άμεσα αλλά και έμεσα από την κοινή γεωργική πολιτική. Ας δούμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά, ας αναλάβουμε δράση όμως το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν, η συνεργασία με τα πανεπιστήμια επίσης, Α μην ξεχνάμε όμω και το ζήτημα τη έρευνα, στο να υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση για την έρευνα. Αυτό όμω δεν μεταφράζεται απαραίτητα πάντα σε περισσότερα διαθέσιμα τρόφιμα. Νομίζω λοιπόν ότι και το ζήτημα των διαθέσιμων τροφίμων θα πρέπει να σε απασχολήσει όπω και οι uh, μικρέ εκμεταλλεύσει. Can... Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ σημαντικό το ερώτημα του πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία τόσων εργασία στις περιοχέ τη Υπέθρου. Από τη δική μου την ε, ιδιαίτερη πατρίδα, εάν αξιοποιούνταν σωστά οι κανόνες της ε, ΚΑΠ, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δημιουργία θέσεων εργασίας και αν είχαν υλοποιηθεί από σχέσεις ε, που είχε δώσει ο Επιτροπός Κάλλας από την κυβέρνησή μας περί της προκαταβολής των ενισχύσεων 11 εκατομμύρια ευρώ θα πέφτανε στην περιοχή σε μικρές εκμεταλλεύσεις όπου και θα δαπανώνταν στη συνέχεια ωστόσο τα χρήματα αυτά δεν δόθηκαν σε ε, μικροκαλλιεργητές αλλά μόνο σε μεγάλους γεωκτήμονες οι οποίοι επίσης όπως και ο μικροκαλλιεργητής, ο μικροκτηνοτρόφος ε, πιάνουν όσο χώρο πιάνει ένα μονό κρεβάτι αλλά τα χρήματα που πήρανε πήγανε όχι στην ε, εκμετάλλευσή τους αλλά σε ένα δεύτερο εξοχικό στην Κροατία και άλλα χού στην Ευρώπη. Εάν λοιπόν θέλετε κάποιε ιδέε για το πώ μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερε θέσει εργασία, το χρήμα τη ΚΑΠ να δαπανάτε στις περιοχές στις οποίες απευθύνεται σε μικρούς γεωκτήμονες. 440 ευρώ ανά άτομο, άντρα, γυναίκα ή παιδί θα αντιστοιχούσαν στη δική μου την περιοχή και από αυτό θα μπορούσαν να προκύψουν πολλέ θέσει εργασία. Ευχαριστώ κύριο Μπράναν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε μια καλή βάση. Ευχαριστώ πολύ τον ε, Ερίκ. Είχαμε μια ομάδα ε, εμπειρογνωμόνων για θέματα της υπαίθρου στη Βόρεια Ιρλανδία που ζητήσαμε να μας δώσουν ιδέες για τις θέσεις εργασίας. 43 ήταν οι προτάσεις τους, σας τις έχω εδώ και θα σας τις δώσω, αλλά πολύ ε, σύντομα να σας δώσω κάποιες ιδέες από, από μια περιοχή νοτιοανατολικής Βρετανίας Βόρειο ανατολικη Βρετανία, συγγνώμη, ε, ε, μας υπόθηκε ότι δεν είναι καλέ οι λύσεις και δεν θα ενισχύσουν την καινοτομία οι επιλογές οι οποίες δείχνουν ιδιαίτερη ε, αποφυγή κινδύνου. Ιδιαίτερα λοιπόν αναφέρονται και σε προγράμματα όπως το Leader που μπορούν να αξιοποιηθούν ως χρήσιμα εργαλεία για την ενίσχυση απασχόληση περιοχές της υπαίθρου, καθιστώντας όμως ταυτόχρονα απολύτω σαφές ότι αυτά πρέπει να ξεκινούν από τη βάση και να μην επιβάλλονται άνωθεν. Μια άλλη σύσταση ήταν πως υπάρχει ο κίνδυνος να προχωρήσουμε ε, λόγω της επιδίωξης όλο και πιο φθηνών τροφίμων και μαζικής παραγωγής σε καταστροφή ουσιαστικά της παραγωγής, προτάσεις σχετικές με τις εκμεταλλεύσεις για την ανάπτυξη της εργασίας, την έρευνα και την ανάπτυξη δηλαδή, που όμως ταυτόχρονα ως έρευνα και ανάπτυξη μπορούν να οδηγήσουν και σε περιορισμό των θέσεων Και βέβαια επιχειρηματικότητα και σχετική κατάρτιση των, κα, των ε, γεωργών και κτηνοτρόφων ήταν πάρα πολύ σημαντική ε, για αυτούς τους ειδικούς της βορειοανατολική ε, Αγγλίας και για το σεμινάριο που κάνουμε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Αλλά θα σας τα δώσω όπω είπα. Ευχαριστώ. Αν ε, μπορούμε να τα βρούμε στο διαδίκτυο, παρακαλώ δώστε μας τις πληροφορίες ή το link για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε όλοι. Ο κύριος Ντές. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ενδιαφέρον όταν συζητάμε το θέμα αυτό και είμαι ευγνώμων για τον συνάδελφο Αντριού, είναι, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ε, Πρέπει πάντα να θυμίζουμε στην κοινή γνώμη ότι ο προπολογισμό της γεωργίας είναι πολύ μικρό ποσοστό, είναι 1% επί του ΑΕΠ, στη δεκαετία του 70-87% και είναι ένας από τους κύριους παράγοντες απασχόλησης η κοινή πολιτική. Το βλέπω αυτό και στη δική μου την ιδιαίτερη πατρίδα, στην ε, Βαβαρία. Έχουμε μπορέσει να συγκρατήσουμε την ανεργία σε πολύ χαμηλά επίπεδα 1,1%, η διπλανή 1,7%, η Βαβαρία όλοι 1,8%. Και εμείς στη Βαβαρία έχουμε και βαριά βιομηχανία. Ωστόσο, η γεωργία είναι ο τομέας με τις περισσότερες θέσεις εργασίας στη Βαταβαρία. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ο δεύτερος πυλώνας και σε αυτό θέλω να πω αγαπητέ συνάδελφε ότι επιτρέπει τα κράτη-μέλη που το επιθυμούν να αξιοποιήσουν συγκεκριμένα κονδύλια της γεωργικής πολιτικής για την απασχόληση. Αυτό έχει μπει σαν λύση. Ξέρω ότι δεν έχει αξιοποιηθεί στη Γαλλία αυτή η δυνατότητα, αλλά ίσως θα ήταν καλό να το κοιτάξετε. Και περιμένω βεβαίως μια περαιτέρω συζήτηση και θα φέρω και εγώ τις δικές μου προτάσεις και τα επιχειρήματα. Ευχαριστώ κυρία Σφένερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον κύριο Αντριέ. Εκ πρώτη το έγγραφο εργασία του αποτελεί ένα εξαιρετικό σημείο αφετηρίας ε, και τροφή για σκέψη για την κοινή γεωρική πολιτική και για το πώς επηρεάζει η κοινή γεωρική πολιτική τι θέση απασχόλησης. Βέβαια, συμμερίζομαι και εγώ τον προβληματισμό των συναδέλφων και διαρωτώ με αν ε, καταφέρουμε να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Αν τα καταφέρουμε και θα βελτιώσουμε την εφαρμογή της κοινή γεωρικής πολιτικής, αλλά και θα θέσουμε τα θεμέλια για μια νέα κοινή γεωρική πολιτική που θα δημιουργεί θέσει απασχόληση. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό το έγγραφο, θα υποβάλω και τροπολογίες, γιατί είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε την πορεία του και πιστεύω ότι έτσι θα συμβάλλουμε στη δημιουργία άμεσων θέσεων απασχόλησης, που δεν θα είναι και επισφαλής ταυτόχρονα και με στο μέσο που θα εξασφαλίσουμε τις άμεσες θέσεις απασχόλησης ε, στην Ήπεθρο ε, θα δημιουργηθούν επαγωγικά και έμεσες θέσεις απασχόλησης. Ναι, ναι, αλλά ε, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης προκαλεί συγκέντρωση στην γεωργία. Γιατί όσο περισσότερο ε, αυξάνεται η συγκέντρωση, τόσο μεγαλύτερη η επιρροή θα έχει η γεωργία. Θα πρέπει όμως να δούμε και την, ε, το συσχετισμό μεταξύ γεωργίας, συγκέντρωσης και οικονομίας. Η κυρία Πετήρ, σας ευχαριστώ. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και χαίρομαι που το εξετάζουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι η γεωργία απορροφά το 40 περίπου το 100 του κοινοτικού προϋπολογισμού. Και με βάση τα στοιχεία που έχουμε, διαπιστώνουμε ότι ε, πάνω από το μισό αυτών των κοινοτικών κονδυλίων προϋπολογισμού ε, πηγαίνουν σε λίγα χέρια, σε πολύ μικρότερο αριθμό γεωργών. Οπότε προσοχή στη συζήτηση θα πρέπει να κατευθύνουμε τους στόχους μας στην ικανοποίηση των αναγκών των οικογενειακών, των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, γιατί αυτές είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινή γεωργικής πολιτικής και θα πρέπει να παραμείνουν στο μέλλον τα θεμέλια αυτής της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και μάλιστα οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις δημιουργούν θέσεις αυτοαπασχόλησης. Εξαιρετικό παράδειγμα και το, από τα καλύτερα παραδείγματα αυτοαπασχόλησης. Πρόκειται για ανθρώπους που δίνουν δουλειά ε, στην οικογένειά τους, που σε καμία περίπτωση δεν είναι... Ε, ε, δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, δεν διεκδικούν επιδόματα ανεργίας, αντίθετα αυτοπασχολούνται και μάλιστα ταυτόχρονα παράγουν τρόφιμα, διαφυλάσσουν την ύπεθρο και προασπίζουν και την, προτε... την ταυτότητα του γεωργικού τοπίου και της ύπεθρου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ε, υπερασπίσουμε αυτές τις ε, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και το μεγαλύτερο τμήμα του γεωργικού προϋπολογισμού θα πρέπει να πηγαίνει στα δικά τους χέρια και όχι στα χέρια των μεγάλων επιχειρήσεων ή των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. που ο μόνος τους στόχος και ο μόνος τους σκοπός είναι να πλουτίσουν. Ευχαριστώ. Κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ πάντως ε, συμφωνώ με το έγγραφο εργασίας ε, του συνέδελφου Eric Καντρέ, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική εργασία εδώ πέρα. Μας δίνει μια καταπληκτική βάση στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε για την επόμενη συζήτηση. Όπως πάνε και οι συνάδελφοι, η κοινή γεωρική πολιτική θα πρέπει να αποτελέσει ένα βιώσιμο πλαίσιο το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει το μέλλον των αγροτικών περιοχών. Επομένω, συμφωνώ πάρα πολύ με τι παρατηρήσει που έκανε ο Ερικ, ιδίω όταν είπε ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε, να επαναπροσεγγίσουμε με διαφορετικό τρόπο την κοινή γεωργική πολιτική, να δούμε πώ θα παράγουμε, με ποιον θα παράγουμε. Ποιε μεθόδους θα χρησιμοποιήσουμε. Αληθεύει το ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν έχει αυτή τη στιγμή ακόμα έναν μετρήσιμο αντίκτυπο όσον αφορά το ζήτημα της απασχόλησης σε αγροτικέ περιοχές. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο και νομίζω ότι η βασική μας εταίροι στα πλαίσια τη γεωργική ανάπτυξη θα πρέπει να δούνε όντω πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα, όπω για παράδειγμα το πρόβλημα τη απασχόληση. Δεν θα ήθελα να, επαναλάβω τις παρατηρήσεις που κάνανε οι συνάδελφοι. Να πω μόνο ότι κάθε φορά που μιλάμε για ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερόμαστε και σε μια νέα γεωργία. Μια νέα γεωργία η οποία θα βασίζεται στην κοινοτομία αλλά και στην απλούστευση του διαδικασιών γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε τελικά να ευνοήσουμε μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη. Σας βλέπω κύριε Πρόεδρε με το σφυράκι και λίγο τρομάζω. θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την προετοιμασία των συνάδελφων, για τη σύνταξη του εγγράφου και τη συνεργασία. Είναι καλό το κείμενο και θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφέρω τη λέξη συγκέντρωση που επισημάνατε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Ναι, η κοινή γεωργική πολιτική ε, κτίνει προς τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας της γεωργικής γης, 3% των επιχειρήσεων της Ευρώπης έχουν 50% της γεωργικής γης στα χέρια τους. Αυτή τη στιγμή, εάν προχωρήσει ακόμη περισσότερο αυτή η τάση, και πάντα η ε, ενίσχυση δίνεται με βάση τις ε, εκτάσεις που έχει κάνει στα χέρια του, τότε ναι θα ενισχυθεί η συγκέντρωση και άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ συγκεκριμένα πού θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσει εργασία, αλλά έχουμε δει ότι η συγκέντρωση γεωργική γη ποτέ δεν γεννά περισσότερε θέσει εργασία. Είναι καλή εκθέση του αδέλφου, πρέπει να την επεξεργαστούμε φυσικά περαιτέρω και θέλω να πω είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο που να νομιμοποιεί την πρόταση αυτή. Γιατί το χρήμα δεν είναι χρήμα του γεωργού, είναι χρήμα τη κοινωνία και ω τέτοιο θα πρέπει να διατίθεται. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριο Άγνιος. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το εξετάσουμε αυτό και υπό τη σκοπιά των φορολογουμένων που χρηματοδοτούν ε, την κοινωνική πολιτική. Τι μπορούμε να περιμένουμε. Έχουμε τους ε, κατοίκους των πόλεων και τους κατοίκους υπαίθρου. Οι κάτοικοι των πόλεων ε, περιμένουν από την κοινή γεωρική πολιτική καλή επιλογή τροφίμων και ποιοτικά τρόφιμα. Αυτά περιμένουν οι κάτοικοι των, φορολογου... οι κάτοικοι των πόλεων και οι φορολογούμενοι που, που χρηματοδοτούν το κοινοτικό προπολογισμό. Βέβαια, στην Ήπεθρο είναι ίσω διαφορετική άποψη. Περιμένουν από την κοινή γεωρική πολιτική περισσότερε θέσει απασχόληση. Βέβαια, με τη μηχανοποίηση που έχουμε, η παραγωγή τροφίμων χρειάζεται λιγότερο κόσμο. Πριν από 50 ε, χρόνια, βέβαια, η απασχόληση στι εκμεταλλεύσει ήταν ε, επώδυνη, κουραστική και βαριά εργασία. Επίσης έχουμε και τα αγροπεριβαλλοντικά συστήματα. Γενικώ πάντως μια κοινή γεωρική πολιτική θα πρέπει να εξαλείπτει τις ε, διακοιμάσεις ε, στην προσφορά και ζήτηση των ε, τροφίμων και των προϊόντων. Τώρα βέβαια έχουμε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, οπότε θέλουμε μια κοινή γεωργική πολιτική που να μειώνει αυτές τις διακοιμάσεις. Βέβαια η δική μου σοβαρή ανησυχία Εντοπίστε στο γεγονός ε, μήπως ε, είμαστε υπερβολικοί στην ε, πιστή και αυστηρή εφαρμογή της ε, πολλαπλού συμμόρφωσης ε, και έχουμε κριτήρια πολύ υπερβολικά. Εμείς ε, βάζουμε 6 δισεκατομμύρια λίρες τερλίνες στην κοινωνική πολιτική και παίρνουμε μόνο 3 δισεκατομμύρια πίσω. Οπότε δεν αρέσει στους Βρετανούς η ιδέα ότι χρηματοδοτούν είτε τις σταυρομαχίες είτε την κτηνοτροφία τάβρων που πηγαίνει στις σταυρομαχίες. Αυτό για εκείνους είναι πραγματικά σκανδαλώδες. Ευχαριστώ κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις παρατηρήσεις. Κανείς δεν μπορεί να έχει αντιρρήσει στη δημιουργία θέσεων εργασία ασφαλώς. Απλώς οι ανταγωνιστικές της εργασία είναι ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί πολύ. Γιατί το να προκύπτουν ε, θέσεις εργασίας οι οποίες όμως δεν επιτρέπουν να επιβιώσει ο εργαζόμενος ίσως δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε. Πολλά μπορούμε να επικρίνουμε σε σχέση με τις προτάσεις, βέβαια, με την ε, ΚΑΠ φυσικά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ολόκληρη, την ευρύτερη εικόνα. Οι άμεσες πληρωμές μπορεί να χρησιμοποιηθούν, δηλαδή να αποδεσμευθούν από το εκτάριο και να πηγαίνουν στον εργαζόμενο, ότι θα του δίνανε 3.500 ευρώ, όχι το μήνα, το χρόνο. Τι θα σήμαινε αυτό, θα ήταν το ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό ε, σε σχέση με την ε, δυνατότητα επιβίωσης σε μια χώρα όπως η Γερμανία επί παραδείγματι και επίσης νομίζω ότι θα ήταν καλό να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία το είπαμε αυτό πρέπει ωστόσο να σημειώνουμε ότι οι θέσει εργασία στον χώρο τη γεωργίας δεν ε, αναπτύσσονται στην, ε, στον πρωτογενή τομέα και αυτό σε ποσοστά 1 προ 8, σε αναλογίε 1 προ 8, 1 προ 10, αλλά σε ε, τομείς σχετικούς με τη μεταποίηση και την περαιτέρω αλυσίδα των γεωργικών προϊόντων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ποιε είναι οι επιπτώσει τη κοινή γεωργική πολιτική στην γαλλική οικονομία. 10 εκατομμύρια ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι απασχολούνταν στο παρελθόν στον τομέα αυτό έχουν μείνει 1 εκατομμύριο, 4% δηλαδή σε σχέση με το 30% που είχαμε στο παρελθόν. Κανένα άλλο οικονομικό κλάδο δεν γνώρισε τέτοια μείωση απασχόληση. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των γαλλικών εκμεταλλεύσεων εξαφανίστηκαν από την δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα και καταλαβαίνετε ότι ο αντίκτυπος ήταν πάρα πολύ αρνητικός στον κοινωνικό ιστό και επαγγελματικό ιστό στις αγροτικές περιοχές. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούμε να σώσουμε τη γεωργία μας και του γεωργού μας αν βγούμε από την κοινή γεωργική αυτή πολιτική, η οποία, όπως σας είπα, κατέστρεψε τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας Είπαμε ότι θα πρέπει καταρχά να έχει την απαραίτητη κυριαρχία κάθε κράτο μέλο, να μπορεί να διαχειρίζεται τι γεωργικέ εκμεταλλεύσει, να μπορεί να επικεντρωθεί πάλι σε εθνικό επίπεδο η παραγωγή, να μπορούν επίση να έχουμε μικρέ μονάδε μεταποίηση σε τοπικό επίπεδο, μονάδε επίση βιολογική παραγωγή. Πρέπει επίσης να δούμε και ποια είναι τα αποτελέσματα των διαφόρων αλλακτικών προϊόντων. Ξέρετε ότι δεν μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε την κοινή γεωργική πολιτική αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι από το 1992 υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα λάβετε όλα αυτά υπόψη, θα κάνουμε πάλι μια συζήτηση άσκοπη χωρίς αυτά τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αλλά το θέμα είναι αν ε, ξεφεύγαμε από την κοινή γεωρική πολιτική, θα είχαμε ε, επιτάχυση τη συγκέντρωση ή, ή όχι. Μάλλον ναι. Ε, Επίση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη μορφή που θα έχει η κοινή γεωρική πολιτική μετά το 2020. Ο κύριο Επιτίδιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, και, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομο. Καταρχά, ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την ε, σημαντική μελέτη που έκανε, την έκθεση που μα παρουσίασε, η οποία καλύπτει πολλού τομεί τη κοινή γεωργική πολιτική και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των γεωργών των χωρών κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δυστυχώ, στα πλαίσια τη κοινή εξωτερική πολιτική και κυρίω τη πολιτική γειτονία δίνουμε τη δυνατότητα σε προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες να κατακλείζουν την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό αφενός με δημιουργεί προβλήματα ασφαλείας γιατί τα προϊόντα αυτά είναι και αμφιβόλου ποιότητας αλλά και κυρίως αμφιβόλου ε, ποιοτικής και υγιεινής ασφαλείας αλλά παράλληλα δημιουργούν συνθήκες αφαιμή του ανταγωνισμού για τα προϊόντα των ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν σαν αποτέλεσμα να ρίχνουν κατακόρυφα τις τιμές των προϊόντων αυτών με αποτέλεσμα και το βιωτικό επίπεδο των γεωργών των κρατών μελών να πέφτει και παράλληλα βεβαίως να μην μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Αυτό το πρόβλημα παρατηρείται κυρίως στους γεωργούς των χωρών του Νότου και πρωτίστως στους γεωργούς της χώρας μου της Ελλάδος, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα δραματικό σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Με πολύ προσοχή διαβάσαμε το έγγραφο εργασία ε, του εισηγητή σα και καταγράψαμε και όλε τι παρατηρήσει κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Ξεκινάει λοιπόν με το έγγραφο αυτό μια συζήτηση για το πώ μπορεί η κοινή γεωργική πολιτική να ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων απασχόληση σε αγροτικέ περιοχέ. Μπορώ να συζητήσω λοιπόν μαζί σα το ζήτημα αυτό. Με πολλού τρόπου η κοινή γεωργική πολιτική μπορεί να οδηγήσει στην βιώσιμη διαχείριση των αγροτικών περιοχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόληση βάσει και των προτεραιοτήτων που ο πρόεδρο Γιούγκερ. Και προφανώ θέλουμε να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τις αγροτικές περιοχές. Περίπου 11 εκατομμύρια αγροτικές εκμεταλλεύσεις δίνουν δουλειά σε 22 εκατομμύρια ανθρώπους και κατά αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν σε αγροτικές περιοχές. Μεταποίηση τροφίμων, πρόθεση τροφίμων, ένας γενικότερος τομέας δημιουργείται που αντιστοιχεί σε 44 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Η κοινή γεωργική πολιτική όμως δεν δημιουργεί μόνο θέσεις απασχόλησης που έχουν σχέση με τη γεωργία. Στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα έχουμε και νέες ευκαιρίες απασχόλησης που έχουν να κάνουν με υποστήριξη προς εταιρείες startups, κάποιες βασικές επενδύσεις ή διάφορες μορφές συνεργασίας και για άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες οι ε, πληρωμές και ενισχύσεις που δίνονται στους ε, γεωργούς δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες προκειμένου να προστατεύουμε το τοπίο, το νερό, το έδαφος. Ξέρετε ότι έχουμε πολλούς νέους γεωργούς οι οποίοι λαμβάνουν υψηλότερε ενισχύσεις. Η ανάπτυξη επίσης ε, της υπαίθρου είναι μια πολύ σημαντική πολιτική που θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πρόκληση τη απασχόληση αλλά και τη οικονομική ανάπτυξη. Πάλι εδώ πέρα μα απασχολεί ιδιαίτερη χρηματοδότηση. Μέσω λοιπόν των προγραμμάτων υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη-μέλη θέλουν να υποστηρίξουν 170.000 νέους γεωργούς, καθώς επίσης και 6.000 νέες start-up μη γεωργικές. Επίσης γίνονται περαιτέρω επενδύσεις προκειμένου να δοθούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης των κλάδων αυτών. Οι δημόσιες επενδύσεις για την περίοδο 2014-2020 για τον τομέα το γεωργικό είναι περίπου 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη προς τις γεωργικές επενδύσεις, προς τους γεωργούς, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεργασίας. Επίσης, ε, υποστήριξη μπορεί να δοθεί μέσω ε, άλλων χρηματοδοτικών μέσων, όπως για παράδειγμα η διακεφάλαια ή η ε, δάνεια και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν και περισσότερα δικά κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν στον τομέα της γεωργίας θα ήθελα να τονίσω ένα νέο στοιχείο στα πλαίσια των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που θα μπορούσε να εμπνεύσει και άλλους τομείς. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης για τη Γεωργία θα στηρίξουμε πάνω από 3.000 καινοτόμα σχέδια όπου θα προσπαθήσουμε να φέρουμε μαζί επιχειρήσεις και κέντρα έρευνα προκειμένου να έχουμε κάποια αυτά αποτελέσματα στον τομέα τη γεωργία. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο την καινοτομία στον τομέα τη γεωργία και κατά αυτόν τον τρόπο τα αποκρινόμαστε στι βασικέ προτεραιότητε έρευνα του προγράμματο Ορίζοντα 2020. Όσον αφορά τώρα τη βιωσιμότητα και την κοινωνική διάσταση. Η βιωσιμότητα μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη χρήση των πόρων. Η κατανόληση πόρων όπω ε, η ηλεκτρική ενέργεια και το νερό είναι σημαντικές προποθέσεις για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Επίσης, ε, μπορεί αυτό να συμβάλλει και στην κυκλική οικονομία και ξέρετε ότι έχουμε και μια δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία. Ένα 51% των, της χρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 14 έως 20 υποστηρίζει περιβαλλοντικά προγράμματα καθώς επίσης και μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Επίσης συμβάλλουμε μέσω των προγραμμάτων αυτών στην προάσπιση των πρώτων υλών της ενέργειας, στην προάσπιση επίσης του αγροτικού τοπίου. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στην γεωργική εκμετάλλευση, αλλά και στην, στα εισοδήματα των γεωργών, καθώς επίσης και στην προστασία του περιβάλλοντος. Θέλουμε να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές και, αυτός, αυτή είναι μια από τις βασικές μας προτεραιότητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις ε, μπορούμε με πιο εύκολο τρόπο στην Ήπεθρο να έχουμε κάποιες, κάποια προγράμματα συνεργασίας ή να προωθήσουμε συνεταιρισμούς. Ένα 54% του αγροτικού πληθυσμού θα καλυφθεί από τέτοιες στρατηγικές πρόθεσης ε, της αγροτικής ανάπτυξης. Θα δημιουργηθούν 44.000 μη γεωργικές θέσεις απασχόλησης και 74.000 θέσεις απασχόλησης που θα έχουν να κάνουν με τον τομέα των υπηρεσιών. Η κοινή γεωργική πολιτική μπορεί να δώσει λοιπόν τη δυνατότητα στον ευρωπαϊκό πληθυσμό να ζει σε αγροτικέ περιοχέ, θα υπάρχει άμεση στήριξη για του ανθρώπου αυτού και θα δημιουργηθούν απαραίτητε προποθέσει για την δημιουργία θέσεων απασχόληση. Θα πρέπει όμω να εκμεταλλευτούμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εφιστάμενα μέσα υποστήριξη που έχουμε. Μολονότι έχουμε πίσω μα 54 χρόνια εφαρμογή τη κοινή γεωργική πολιτική, υπάρχουν πάρα πολλοί που θεωρούν ότι η κοινή γεωργική πολιτική εξακολουθεί και έχει μια σημαντική προστιθέμενη αξία. Το αυτό και στην τελευταία δημοσκόπηση που έγινε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε ποιε είναι οι δυνατότητε απασχόληση προσφέρει η κοινή γεωργική πολιτική και προσβλέπουμε και στην περαιτέρω συνεργασία που θα έχουμε μαζί σα στα πλαίσια τη έκθεση αυτή. Σας ευχαριστούμε. Ο εισηγητής μας τώρα, ο κύριος Αντριέ Παρακαλώ, θα θέλετε να σχολιάσετε τις παρατηρήσεις των συναδέλφων μετά από την πολύ καρποφόρα συζήτηση. Να σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και όλους τους συναδέλφους για τις τοποθετήσεις τους. Πολύ ενδιαφέρουσες όλες και πολύ πλούσιες. Είναι ακριβώς άλλωστε αυτός και ο στόχος αυτής της πρώτης ανταλλαγής απόψεων, να επαναπροσδιοριστεί δηλαδή το πλαίσιο, το συγκεκριμένο πλαίσιο της εκθέσεως. Θα είδατε ότι το έγγραφο αυτό δεν περιορίζεται στην ε, ανάπτυξη του περιεχομένου της εκθέσεως, αλλά αντιθέτως κάπως προκλητικά θα έλεγα να θέσει ζητήματα και να πλαισιώσει μελλοντικές προτάσεις. Ξεκινώ από τις τοποθετήσεις τη Επιτροπής. Την απάντησή μου γιατί από αυτά που μας λέτε δεν έχει λόγο ύπαρξη αυτά η έκθεση. Πάνε όλα πολύ καλά, δεν υπάρχει λόγος να διερωτηθούμε ε, πώς πάει αυτή η μεταρρύθμιση, γιατί ο κόσμος είναι όμορφος και αγγελικά πλασμένος. Αυτό μου λέτε. Πάντως, όποιος ε, αντιμετωπίζει την πραγματικότητα στις περιοχές της υπαίθρου, βλέπει πολύ καλά ότι αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Εγώ βλέπω τα προβλήματα που έχουν ε, οι ε, εκτροφή στη Βρετάνη της Γαλλίας, η Γεωργία, γενικότερα προβλήματα που ανέφεραν και οι συνάδελφοι. Είναι πολλά τα προβλήματα λοιπόν που εντοπίζονται στην πραγματική ζωή και ερωτηματικά που έχουν να κάνουν με το μέλλον. Άρα ναι, τα βραχυπρόθεσμα πρέπει να τα δούμε, αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να αποκλείουμε και τη συζήτηση για τη μέσο πρόθεσμη προοπτική. Και αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, μια και το, αναφέρατε και το ανέφερα και εγώ στην αρχική μου τοποθέτηση, το θέμα της συγκέντρωσης πρέπει να δοθούν από την έκθεση συγκεκριμένε απαντήσεις ναι, ασφαλώς, αλλά δεν μπορούμε και να μην διερωτηθούμε για τα θέματα ουσίας, τα θεμελιώδη ζητήματα. Μια δημόσια πολιτική, κρατική πολιτική δεν θα πρέπει να συνοδεύει κάθε γεωργικό πρότυπο με την υποστήριξή της ή όχι. Δεν πρέπει να μας απασχολεί στο ζήτημα. Η πολιτική για την Ήπειθρο, για τη Γεωργία δεν έχει συνέπειες σε κάθε σημείο της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από το ερώτημα. Έχουμε ε, ερωτηματικά που προκύπτουν ακόμη και σε σχέση με την ανάπτυξη μιας γεωργικής παραγωγής στα αστικά κέντρα. Ε, η διάχυση των θέσεων εργασίας μέσα σε διαφορετικές χωρικές ενότητες έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης. Άρα λοιπόν ε, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι η γεωφυσική συνθήκη, δηλαδή πρόκειται για πεδιάδα, πρόκειται για ορεινή περιοχή, πρόκειται για απομακρυσμένη περιοχή και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Πολλά χρόνια τώρα διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά αποζημιώνουμε την απώλεια οικονομικής δραστηριότητας από τη γη μας με τις ενισχύσεις. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε και τις προτάσεις των, αλλά και τις μελλοντική, ή πάνω απ' όλα της μελλοντική. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό οπλοστάσιο που θα πρέπει για τα επόμενα χρόνια να ξανασχεδιάσουμε και για την κυρία Εράνς Καρσία ασφαλώς το θέμα δεν είναι να κάνουμε ε, σχεδιασμό κήπων αλλά γεωργική οικονομία. Μιλήσατε κι εσείς για ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Πρέπει να κοιτάξουμε να δουλέψουμε αυτόν πόρο που ονομάζεται έδαφος χωρίς να τον καταστρέφουμε. Είναι αυτό ένα κύριο διακύβευμα. Το έδαφος είναι και στην ανάπτυξη βασικός πόρος. Το ίδιο ισχύει και για το νερό, το ίδιο ισχύει για τον ατμοσφαιρικό αέρα. Στη γεωργία λοιπόν όλα αυτά συνδυάζονται. Είναι μεν καθήκον πρωταρχικό της γεωργίας η παραγωγή τροφίμου, αλλά έχει μια πολύ ευρύτερη λειτουργία ως προς τη διαφύλαξη οικοσυστημάτων και περιβάλλοντος. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια. Σημειώνω κύριε Πρόεδρε τις παρατηρήσεις σας για την πλαισίωση της δουλειάς μου στο μέλλον. Με μεγάλη χαρά θα σας παρουσιάσω τις επόμενες προτάσεις και βέβαια θα συνεργαστούμε από σήμερα εντατικά με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ήταν ε, έγγραφο εργασία αυτό που μα έχετε υποβάλει μέχρι στιγμή και αυτή ήταν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Σίγουρα με την όλη συζήτηση θα εμπλουτιστεί η γνωμοδότηση αυτή και θα συνεχιστεί η συζήτηση στις 25 και 26 Απριλίου που θα γίνει και παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. έχουμε αρκετό καιρό μέχρι τότε. Οπότε ολοκληρώνουμε το σημείο 8 και γυρίζουμε στο προηγούμενο, στο σημείο 7, τη νέα συμμαχία για την επιχειριστική ασφάλεια και τη διατροφή. Όπως σας είπα, γνωμοδότηση θα συντάξουμε, γιατί επί της ουσίας είναι αρμόδια η Επιτροπή ΔΕΒΕ. Η συντάκτρια γνωμοδότηση Επιτροπής Γεωργίας είναι η κυρία Μόλι Σκοτ Κάτω. και μιλούμε για την ε, νέα συμμαχία που γίνεται από τον προηγούμενο Μάιο και γίνεται πρόταση για αύξηση των ιδιωτικών και των δίωμασων επενδύσεων προκειμένου να ισχυθεί η γεωργία και να ληφθεί υπόψη ο, ο ρόλος της γεωργίας ε, και της παραγωγής τροφίμων. Όπως σας είπα, θα συντάξουμε γνωμοδότηση. Αρμόδια εισηγήτρια, συντάκτρια είναι η κυρία Σκοτκάτο, στην οποία και δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ μαζί σας ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα ε, ζητήσαμε τη γνώμη και εμπειρογνωμόνων κατά τη σύνταξη της γνωμοδότησης. Γνωρίζετε τον Άλμπερτ Σούτερ, που είναι, ήταν ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στα τρόφιμα. Και μάλιστα στην έκθεσή του για την ε, νέα αυτή συμμαχία ε, μιλάει για το ε, απαρχημένο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε μέχρι στιγμή για τη Γεωργία. Σε ό,τι αφορά τον τίτλο αυτή τη οργάνωση, ε, φυσικά μιλάει για την διατροφή, αλλά δεν αρκεί να περιοριζόμαστε στη διατροφή. Η διατροφή είναι δευτερεύον θέμα για τις ε, ευκαιρίες που δίνει ο αγροπιστικός τομέας. Δεν δίνεται έμφαση στα υγιεινά τρόφιμα, αλλά περισσότερο στα γεωργικά προϊόντα. Κάτι που πιστεύουμε θα αυξήσει την ε, εξάρτησή μας από τη γη και την... το πρόβλημα που δημιουργεί η διάβρωση και η υποβάθμιση του, του εδάφους. Ελπίζω η Επιτροπή Ανάπτυξης να λάβει υπόψη τις ανησυχίες της ε, κοινότητας αναπτυσσομένων χωρών. Ε, έχουμε λάβει έγγραφα από πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, από την Global Justice Now, την Action Aid, την Γαλλική Οργάνωση Action Against Hunger, την, το, Αφρικανικό Κέντρο για την Βιοασφάλεια, την Oxfam και άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις που επεσήμαναν τις αδυναμίες και τις αποτυχίες αυτής της για να σα δώσω ένα παράδειγμα που μα έδωσε η Global Justice Now. Ε, στην πολιτεία Ταράμπα τη Νιγηρίας, μια παραχώρηση 30.000 νεκταρίων ε, δόθηκε σε μια αμερικανική εταιρεία για να ξεκινήσει η οριζοκαλλιέργεια, χωρί όμω προηγούμενη διαβούλευση τη το, το, τοπικής κοινότητας ε, και των 40.000 ανθρώπων που εξαρτώνται από τι καλλιέργειε αυτέ για το βιοπορισμό του. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι τι κάνουν, αλλά εγώ λαμβάνω χιλιάδε επιστολέ. 500 ε, μόνο την περασμένη εβδομάδα ε, με ανησυχίες των πολιτών για το έργο αυτής της νέας συμμαχίας. Τι κάνει λοιπόν η γνωμοδότηση. Μας ενδιαφέρει μια ανθεκτική ε, εγχώρια παραγωγή τροφίμων. Είναι σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές στην αγορά και κυρίως να αντιμετωπίσουμε και τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, να ενθαρρύνουμε μεγάλη ποικιλία, μεγαλύτερη ποικιλία απορροκυπευτικών για να βελτιώσουμε τη διατροφή μα. Επίση, οι πολιτικέ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη συμμετοχή των γυναικών και των μικρών καλλιεργητών. Αυτέ θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο τη πολιτική μα, γιατί είναι και η πλειοψηφία των γεωργών στον κόσμο. Επίση, ε, η πρωτοβουλία που εξετάζουμε θα πρέπει να ε, επιτρέψει στους γεωργούς ε, να αποφύγουν την αλληλεξάρτηση. Δεν μπορούμε ε, να έχουμε υγιεινά τρόφιμα αν οι γεωργοί είναι συνεχώς εξαρτημένοι αυτό το φαύλο κύκλο των ε, φυτοφαρμάκων, ε, των λιπασμάτων και του εδάφους. Θα πρέπει να προωθήσουμε την αγροβιοπικιλότητα με τοπικές τράπεζες σπόρων και πρόθεση των γηγενών σπόρων. στο θέμα της αρπαγής της γης, ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που ενδιαφέρει και τη Νέα Συμμαχία υπάρχουν ε, προφανή φαινόμενα και κερδοσκοπίες και ε, ε, απατών και κυρίως η αρπαγή των γεών ε, εστερεί από τους μικροκαλλιεργητές βασικούς, βασικές πηγές βιοπορισμού. Άλλα θέματα που ενδιαφέρουν κυρίως τους Ευρωπαίους Γεωργούς είναι οι ασθενείς θέσεις τους στις διαπραγματεύσεις, η μικρή αθάριση που γίνεται στις, στην παραγωγών και η ελάχιστη διαπραγματευτική ισχύ που έχουν στην επιστηστική αλυσίδα. Αν εφαρμόσουμε διεθνεί προδιαγραφέ όπω είναι τα ε, οι προδιαγραφέ τη ΦΑΟ ή του Ηνωμένου Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, θα πρέπει ε, να διαπιστώσουμε ότι οι φτωχότερε τη αναπτυσσόμενε χώρε δεν συμμερίζονται τι δικέ μα ανησυχίε και προβληματισμού. Ευχαριστώ του και ηγητέ για τα σχόλια του και προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία για να καταλήξουμε σε γνωμοδότηση που θα τύχει ευρεία υποστήριξη στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα κατακλείδη να πω ότι ε, ζητούμενο είναι ε, μια νέα συμμαχία που θα εξασφαλίσει πραγματικά την επιστηστική ασφάλεια και τη διατροφή, αλλά δεν θα διακυβεύσει τη δυνατότητα των φτωχότερων συμπολιτών μας ε, να παράγουν αρκετά τρόφιμα ώστε να μπορούν να εξασφαλίζουν τη διατροφή τους και το βιοπορισμό τους. Ευχαριστώ. Κύριε you, um, uh, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω απολύτως μετά όσο μας είπε η Μόλη. Όντως, η προσέγγισή μας είναι ιδιαίτερα παροχημένη και τα πράγματα πολλές φορές είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ακούσαμε. Ξέρετε ότι εργάστηκα στον τομέα της Αναπτυξιακή βοήθειας ε, στα πλαίσια της Christian Aid στο παρελθόν πρωτού γίνω Ευρωβουλευτής ε, και πολύ σαν γνωρίζουμε ότι η απάντηση στην παγκόσμια ένδια, στην παγκόσμια πείνα δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Αντίθετα έχει να κάνει με τα οικονομικά συστήματα τα οποία ισχύουν. Ξέρετε ότι πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν με τα κονδύλια και τα χρήματα, αλλά τα χρήματα έχουν να κάνουν τελικά με φιλανθρωπία και στην πράξη δεν τροποποιούν τους βασικούς διαρθρωτικούς λόγους της φτώχειας. Δεν μπορεί να αποτελέσει σε καμία περίπτωση λοιπόν πανάκια η χρηματοδότηση. Αντίθετα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια τα οποία έγκυται, έγκυται τελικά στα οικονομικά συστήματα τα οποία ακολουθούμε αλλά και σε άλλα ζητήματα όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια πείνα και την παγκόσμια φτώχεια στο παρελθόν κυρίως μέσω της αντιξιακής βοήθειας και μέσω της αντιμετώπισης του χρέους του τρίτου κόσμου, όπως λέγαμε στο παρελθόν. Το ότι καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε το αθέμητο διεθνές εμπόριο και το ότι καταφέραμε να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε επίση και το ζήτημα τη φοροδιαφυγή ή τη αποφυγή καταβολή φόρων, τόσο στο νότιο όσο και στο βόρειο ημισφαίριο. Και αυτό το οποίο βλέπουμε ως προ αυτό είναι ότι ορισμένε επιχειρήσει, ε, οι οποίε φαίνεται ότι συμμετέχουν σε αυτή τη νέα συμμαχία για την επιστηστική ασφάλεια και την διατροφή, είναι τελικά πολύεθνικέ, ε, οι οποίε έχουν εξειδικευτεί εντό αγωγικών στην αποφυγή καταβολής φορολογικών εισφορών και μάλιστα το κάνουν αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξέρετε λοιπόν ότι από τη μία πλευρά έχετε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες εμφανίζονται εδώ πέρα ως οργανισμοί οι οποίοι υποστηρίζουν τη σχετική αυτή πρωτοβουλία αλλά εγώ γνωρίζω στην πράξη ότι πολύ συχνά φοροδιαφεύγουν και κατά αυτόν τον τρόπο δεν δίνουν τη δυνατότητα σε αφρικανικές χώρες να έχουν πρόσβαση σε εκατομμύρια και εκατομμύρια δολάρια, το οποίο είναι ένα απολεσθέν κέρδος για τις χώρες αυτές και ανταυτού τελικά τους δίνουν μερικές χιλιάδες δολάρια ως αναπτυξιακή βοήθεια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο και θα έλεγα και εντελώς εσφαλμένο από ηθικής πλευράς. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που μπορώ να συνεργαστώ για το ζήτημα αυτό με τη Μόλη. Μα είπε ότι όντω υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία λείπουν από την προσέγγιση αυτή. Μια σημαντική απουσία είναι αυτή τη κοινωνία των πολιτών. Πρέπει και η κοινωνία των πολιτών να εμπλέκεται περισσότερο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε επίση το ζήτημα τη αρπαγή τη γη, το ζήτημα τη ιδιωτικοποίηση του τομέα των σπόρων, το ζήτημα των εξαγωγών, ενώ θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο το διαπεριφερειακό εμπόριο. Και επίσης δεν αναφερόμαστε καθόλου εδώ πέρα στην διάσταση του φύλου, γιατί όπως ακούσαμε και στην Αφρική αλλά και γενικότερα στον αφισόμενο κόσμο οι περισσότεροι γεωργοί είναι γυναίκες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε επίσης και στον αγρο... αγροδασοκομικό τομέα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να συνεργαστούμε αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της έκθεσης αυτής αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρουμε να οδηγηθούμε σε πολύ θετικά αποτελέσματα τη στιγμή που οι βάσει από την οποία ξεκινάμε είναι αρκετά σαφροί. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να μην ξεπερνάτε το χρόνο σα. Η κυρία Ριμπέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συντάκτηρα γνωμοδότηση για την πολύ σημαντική αυτή γνωμοδότηση. Ε, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2012 με διεθνείς εταίρους και στόχο ε, να βγουν πολλές χώρες, ιδιαίτερα της υποσαχάριου Αφρικής, από το πρόβλημα της, ε, του λοιμού που αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει να γίνει συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για τη βελτίωση της γεωργίας και του αγροπιστικού τομέα 10 αφρικανικών χωρών. Ε, βέβαια, έκανα μία ε, έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών και βρήκα κάποιες πολύ επικριτικές θέσεις για την αυτή συμμαχία. Μερικοί τη χαρακτήρισαν και νεοεπικιοκρατική προσπάθεια. Αναφέρθηκε το θέμα της αρπαγής ε, των εδαφών, των γεών, του, του νερού και άλλων ε, φυσικών πόρων. Ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα όμως με τόσο ευγενείς στόχους δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζει τόσο ανησυχητικά. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο πώς θα ευθυγραμμίσουμε αυτό το πρόγραμμα με τους αρχικούς του στόχους, ώστε να ωφελήσει τους πραγματικούς δικαιούχους. Τι φτωχέ και αναπτυσσόμενε χώρε. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι θα πρέπει να επαναπροσυνατολίσουν το στόχο το, της Νέας ε, στην, ε, στη βασική γεωργία βιοπορισμού και φυσικά να ενθαρρυνθούν οι οργανώσει των παραγωγών και οι συνεταιρισμοί για να ενισχυθεί η διαπραγματευτική του ισχύ. Επίση, ε, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη βιοπικιλότητα, ε, και στην, ε, ε, καλύτερη θέση των οργανώσεων παραγωγών στις διαπραγματεύσεις. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε και την ισότητα των δύο φύλων. Θα πρέπει να ληφθεί και αυτή η υπόψη και καλό θα ήταν να παρατείνουμε το, πρόβλημα, το πρόγραμμα και σε άλλες αφρικανικές χώρες που έχουν σημαντικές ε, μεταναστευτικές ε, ροές και αντιμετωπίζουν δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση εξαιτίας ε, της έλλειψης τροφίμων ή της υπερεκμετάλλευσης των γεών. Ευχαριστώ και με στη διάθεσή σας για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ κύριο Σαντριού. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την κυρία Γουλσκουτ Κάτω για την έκθεσή της και να της πω ότι υποστηρίζω και συμμερίζομαι την προσέγγιση της. Η υποστήριξη της γεωργίας και της υπαίθρου πάνω απ' όλα σημαίνει αλληλεγγύη. Να βοηθούμε αυτούς που πλήττονται από λοιμό. Μέχρι και 80% από αυτούς οι οποίοι υποσυτίζονται στη σημερινή εποχή και είναι παράδεξο είναι γεωργοί. Δεν έχουν δηλαδή επαρκείς πόρους παραγωγής. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες, περιοχές στον κόσμο όπου επιχειρήσεις, κερδοσκόποι, άλλες δυνάμεις έχουν στα χέρια τους την εκμετάλλευση της γης. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε αυτό υπόψη στην πολιτική της αναπτυξιακής συνεργασίας. Στον αγώνα για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής κρύβονται και σημαντικές γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις, νέες πολιτικές ε, μεταναστευτικές ροές, πρόσφυγες για λόγους κλιματικών αλλαγών. Είναι όλα ζητήματα που πρέπει να κοιτάξουμε και πρέπει να αλλάξει ένα πρότυπο παραγωγής με τη βιοπικιλότητα, με κατάλληλες ανάλογα με το οικοσύστημα μεθόδους παραγωγής, εναλλαγή, όχι μόνο καλλιέργεια και αυτά, Πρόεδρε, είχα να πω εγώ για να ενισχύσω, για να δώσω τροφή συζήτηση και να υποστήριξω για άλλη μια φορά την πρόταση της συναδέλφου. Αγνιού. Ε, ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο πρόσφατα κάλυψα και βρίσκω πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η Γερμανία σε αξία εξάγει περισσότερο κατεργασμένο καφέ από ότι ολόκληρη η Αφρικανική Ήπειρος σε ακατέργαστο καφέ. Προφανώς δεν πρόκειται για καφέ ο οποίος τροφοδοτεί μόνο την ευρωπαϊκή αγορά, άρα δεν είναι ε, προς όφελος του Ευρωπαίου Γεωργού αυτή η ανταγωνιστική σχέση με τον Αφρικανό ε, καφέ, καφέ καλλιεργητή. Γιατί λοιπόν να μην μειώσουμε τους δασμούς στον καφέ. Επίσης αποτυχίες της ε, γεωργίας της Αφρικής είναι αποτυχίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξάρτηση από την ε, συντήρηση που μπορεί να προσφέρουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στη γεωργία αυτή αλλά και στη Βρετανία συμβαίνει το ίδιο και δεν είδα να μας προβληματίζει, να μας προξενεί δυσκολία το γεγονός ότι είμαστε εξαρτημένοι από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αντιθέτως, μάλιστα, και βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, πολύ συντηρητική σχέση, ε, ε, έχει πολύ συντηρητική θέση για τα γενετικά τροπημένα προϊόντα και σε αυτό κάνει πολύ μεγάλο κακό στην Αφρική και μπορεί να καταλήξει ακόμη και σε διάβρος των εδαφών, να καταλήξουν μεγάλες περιοχές της Αφρικής γιατί δεν επιτρέπει να φυτευθούν γενετικά τροπημένοι οργανισμοί. Να σας πω τι προϊόντα μπορεί να υπάρχουν στην Αφρική. Ξέρω ότι ο καπνός δεν είναι τροφή. Μεγάλε ήταν οι εκμεταλλεύσει που καλλιεργούσαν καπνό. Έχουν φύγει όλοι αυτοί οι καλλιεργητές. Τώρα είναι μικρότεροι καλλιεργητέ, Αλλά η απαγόρευση χρήση προϊόντων καπνού ε, οι περιορισμοί τέλο πάντων είναι ει βάρο των παραγωγών. Αυτοί οι Αφρικανοί λοιπόν καλλιεργητές της Ζιμπάουμπουε εξαρτώνται απολύτω από τις επιδοτήσεις για την επιβίωσή τους. Επίσης, Ε, αντί να επιτραπεί ε, στην, ε, στους χωρικούς να φωνεύουν μόνο τους τις λεοπαρδάλεις οι οποίες καταστρέφουν τις, την κτηνοτροφική τους παραγωγή γιατί σκοτώνουν τα ζώα τους θα έπρεπε να το λένε στις αρχές, οι αρχές να καλούν πλούσιους Αμερικανούς θα πληρώνουν και πολλά λεφτά για το σαφάρι αυτό έτσι θέλανε τα προβλήματά τους Ο κύριος θα πρέπει σίγουρα να στηρίξουμε τη τοπική και εθνική παραγωγή. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει και τη βάση τη γεωργική πολιτική. Αυτό ήταν το ζητούμενο για όλου. Δυστυχώ όμω αυτό το σχέδιο δεν αφορά του Ευρωπαίου γεωργού. Για τι αναπτυσσόμενε χώρε η γεωργία είναι ένα τρόπο για να στρέψουν τον πληθυσμό του και να σταθεροποιηθούν γεωγραφικά. Με την διαιώνιση τη εξάρτηση θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε τίποτε στι αναπτυσσόμενε χώρε, αλλά να σεβαστούμε τι γνώσει του και τι τοπικέ παραδόσει. Έχω πολλέ αμφιβολίες όμως και πολλούς φόβους. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μελέτες να μας εξηγήσει με ποιο τρόπο θα ενθαρρύνει σταθερές παραγωγές ικανές να θρέψουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Γιατί μόνο δήλωση προθέσεων έχουμε μέχρι στιγμής. Γιατί καταγγέλλεται κάποιε ροέ. Αν σταματήσουμε τη συγκέντρωση των εκμεταλλεύσεων σε λίγα χέρια, ώστε να δώσουμε έφαση περισσότερο σε παραδοσιακή γεωργία, τότε θα πρέπει να αλλάξουμε το σύστημά μα. Είναι μια διαφορετική γεωργία αυτή. Δεν είμαι κατά, αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο, γιατί τελικά δεν ξέρουμε πού το πάτε. Θέλετε μια παραδοσιακή γεωργία μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων ή μια βιομηχανοποιημένη γεωργία με μεγάλες εκμεταλλεύσεις που θα προσανατολίζεται στις εξαγωγές. Θέλετε βιομηχανικές χώρες μεγάλων καλλιεργειών και αναπτυσσόμενες χώρες με παραδοσιακή γεωργία μικρή εμβέλειας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. κυρία Μίλλερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα στην εισηγήτρια. Είναι μια καλή ε, τοποθέτηση με ένα πολιτικό μήνυμα. Χρειάζεται μια νέα συμμαχία για την επιστηστική ασφάλεια. Πρέπει αυτή τη συμμαχία να τη δημιουργήσουμε. Σημαντικό, απαραίτητο, είναι ο μέσο και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την γεωργική οικονομία, την επιστηστική ασφάλεια να προχωρήσει. Ο έλεγχος από πλευρά των ε, αλλοδαπών επενδυτών πρέπει να σταματήσει και βέβαια είναι κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη αυτών των φτωχών περιοχών της υπαίθρου. Οι γυναίκες, η μεταφορά της γνώσης και τεχνογνωσίας είναι νομίζω κύρια καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να προσφέρουμε βοήθεια για διεθνείς ανταλλαγές ιδιαίτερα στο τομέα της γεωργικής καλλιέργειας. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε καλή εμπειρία από αναπτυξιακή βοήθεια. Έχουμε παραδείγματι την εταιρεία διεθνούς συνεργασίας όπως λέγεται στη Γερμανία, γνωστός παλαιός και αποδεδειγμένα καλός εταίρος και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Κύριε Σταγαμπηλά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θα σας κρατήσω πολύ. Θέλω να συνοψίσω μόνο εκ μέρους ομάδας τη θέση μας σχέση με την έκθεση της συναδέλφου. Πολύ μεγάλη ποιότητά της, πολύ καλό το περιεχόμενό της. Μόνο στο σημείο είναι εκεί που μιλάει για την εθνική μιλάει για εθνική παραγωγή τροφίμων, επειδή η Ευρώπη δεν είναι έθνος, καλό θα είναι να μιλάμε για χώρια ή εσωτερική Πάντως το πνεύμα είναι σωστό, δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα και ζητώντα το λόγο νομίζοντα ότι ο Πολ ε, Μπραν πολύ σωστά συνόψισε τις θέσει μας, ε, αρκούμε σε αυτά τα ολίγα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Φλάνναγκαν. Ευχαριστώ. Ε, με κάλυψαν οι προλαλήσαντε σε μεγάλο βαθμό. Ε, συμφωνώ με τη Μόλη και στηρίζω το έργο της. Κάθε μέρα όταν έρχομαι στην Επιτροπή ακούω πώς θα θρέψουμε τον κόσμο. Αλλά βρίσκομαι ως ε, άθεος ε, σε δύσκολη θέση γιατί θα πρέπει να σας υπενθυμίσω τη βίβλο που λέει ε, δεν χρειάζεται να θρέψουμε εδώ. Ε, δώσε ένα ψάρι στον άλλον και θα τον ε, θρέψει για μία μέρα. Αν του μάθει να ψαρεύει, θα τον θρέψει για μια ζωή. Βέβαια, εντάξει, αυτά ακούγονται λίγο σαν κήρυγμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ε, τι ευκαιρίε για τον βιοπορισμό στου Γεωργού. Ο κ. Δέσ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την ε, η συγγήτρια υποστηρίζω τα είπε ο προλαλή σα την αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να αναλογιστούμε εκ βάθρων τα πάντα. Είχα τη δεκαετία του 80 μια ιδιωτική πρωτοβουλία με ένα σχέδιο στην Βραζιλία όπου υπάρχουν και πολλοί μικροπαραγωγοί οι οποίοι δεν έχουν αρκετό, αρκετή τροφή για να ε, καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Είχαμε λοιπόν κάνει μια ε, μεγάλη προσπάθεια με έρανο για να μαζέψουμε χρήματα και έτσι αγοράσαμε αγελάδα που την δανείσαμε στον παραγωγό. Τη δανείσαμε, δεν την πουλήσαμε, ούτε τη χαρίσαμε. Ε, με τον όρο ότι μπορούσε το πρώτο χαράκι να το κρατήσει για δικό του, το επόμενο όμως θα έπρεπε να μας το επιστρέψει. Και έτσι λειτουργήσε αυτό το σχέδιο. Υπάρχουν πολλά άλλα, εκατοντάδες μπορώ να σας αναφέρω. Και ο κύριος Αντριέ είπε πολύ σωστά ότι είναι 80% από αυτούς που λιμοκτονούν παραγωγή γεωργική. Έχουμε τώρα μάλιστα έναν συνάδελφο από τον Bundestag της Γερμανίας, ο οποίος είναι στην Αιθιοπία για να βοηθήσει μικρούς παραγωγούς να αναπτύξουν την παραγωγή τους κατά τρόπον ώστε να μπορούν τουλάχιστον να θρέφουν τις οικογένειές τους. Είναι καλύτερο να στρέψουμε το βλέμμα λοιπόν προς τα μικρότερα έργα και project. Τα μεγάλα δεν, ε, για τα μεγάλα δεν έχω μεγάλη εκτίμηση. Άλλωστε όταν έχουμε να κάνουμε είτε με δικτατορικά καθεστώτα είτε με εκτάσεις, δυστυχώς την κυρία Νόχλη δεν την ακούσαμε, ε, είτε με εκτάσεις εκατομμυρίων τετραγωνικών ε, που ανήκουν σε Κινέζους στις χώρες αυτές, τα μεγάλα project δεν είναι χρήσιμα. Πρέπει να κοιτάξουμε μικρές λύσεις και να προσέχουμε τα δικτατορικά καθεστώτα που συμβαίνει στη Ζιμπάμπουε να μην οδηγούν σε επισητιστικό κίνδυνο, σε λοιμό τους ίδιους τους πληθυσμούς απαγορεύοντας την παράδοση της ευρωπαϊκής βοήθειας. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε είναι σημαντικό να φροντίσουμε για την επιθετιστική ασφάλεια παντού στον πλανήτη. Και φυσικά δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε τι γίνεται με τη μεταναστευτική κρίση και τι θα συμβεί σε περίπτωση που κάποιες, σε κάποιες περιφέρειες της χώρας τα πράγματα παίρνουν διαφορετική τροπή από ό,τι περιμέναμε. Ήδη έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες και νομίζω ότι είναι κάτι που αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη και να επικρίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εμπλακεί στην πολιτική αυτή για να προωθήσει την επιστημιστική ασφάλεια στις χώρες αυτές. Επίσης η συζήτηση μας δίνει μια μεγάλη ευκαιρία να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγήσει και λεπτομέρειες τι γίνεται με αυτό το φαινόμενο της ε, αρπαγής των γεών. Ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάποια τέτοια κρούσματα. Θυμάμαι ότι τα έχουμε συζητήσει και στην Επιτροπή. Σε μερικές χώρες, ιδιαίτερα της Ανατολικής Ευρώπης, υπάρχει πρόβλημα με την αρπαγή των γεών. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, 43% των γεωργικών εκτάσεων στη Ρουμανία βρίσκονται ε, στα χέρια τριών, τεσσάρων μεγάλων ομίλων, εταιριών ή μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων ή νομικών οντοτήτων. Και μάλιστα αυτές οι νομικές οντότητες, ε, μια και έχουν τίτλους ιδιοκτησίας για τις διαρκές αυτές εκτάσεις, είναι, ε, έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν για το, τη χρήση τους. Κάτι που μπορεί να δημιουργήσει τεράστια ανισορροπία στην Ρουμανική Γεωργία, παράδειγμα. Θα πρέπει και αυτό το φερόμενο να το λάβουμε υπόψη που λαμβάνει χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Σλάιερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος ε, Μπούντα με πρόλαβε. Και είπα αυτά που ήθελα να πω εγώ. Η μεταναστευτική κρίση θα πρέπει να μας κινητοποιήσει, γιατί βλέπουμε τι προβλήματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον. Ε, κοιτάξτε την Κίνα, τις ασιατικές χώρες, ε, τι συμβαίνει εκεί. Δεν πρέπει να υποτιμούμε το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Εξαντλήθηκε ο κατάλογος των αγορητών. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Σκοτ Κάτο, για να δευτερολογήσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τη θετική αυτή συμβολή πολλών ομιλητών και για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση που είχαμε σήμερα το απόγευμα. Όσον αφορά τις τροπολογίες, Νομίζω ότι πρέπει σαφώς να συζητήσουμε το ζήτημα της βιωσιμότητας των γεωργών, το ζήτημα των επιδοτήσεων. Ξέρετε ότι δεν μπορούν πάρα πολλοί γεωργοί να αγοράζουν τις σημαντικές πρώτες λύσεις, ύλες τις οποίες χρειάζονται. Επίσης, χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα. Θα ήθελα να λάβουμε υπόψη μα τι ε, ιδέε του Πολ. Ο Πολ αναφέρθηκε επίση σε διάφορε επιχειρήσει οι οποίε αποφεύγουν να καταβάλουν ε, φορολογικέ εισφορέ και κατά αυτόν τον τρόπο δεν δίνουν το απαραίτητο εισόδημα ή τα απαραίτητα χρήματα στι πιο φτωχέ χώρε. Ξέρετε ότι ε, Μία από τις τροπολογίες που είχαμε καταθέσει προς την έκθεση DOTS ήταν σχετική με αυτό το ζήτημα, δηλαδή να καταφέρνουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσαμε δεχομένως και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας στα πλαίσια της νέας αυτής συμμαχίας και δεν μπορώ να δεχθώ όμως κάποιες τροπολογίες που θα έχουν να κάνουν με το κυνήγι σε χώρες της Αφρικής. Βασικός στόχος είναι εδώ πέρα να προασπίσουμε τους πιο φτωχούς, να καταφέρουμε επίσης να δίνουμε την απαραίτητη ποσότητα τροφίμων σε όλους τους ανθρώπους στις χώρες αυτές, ότι δραστηριοποιεί τη συμμαχία. Ευχαριστώ. Μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου έχετε δύο για την υποβολή τροπολογιών. Ευχαριστώ την συντάκτρια γνωμοδότηση, την κυρία Μόλι Σκοτ Κάτω και περνούμε στο προηγούμενο σημείο, το παίρνουμε το σημείο 6, τις τεχνολογικές λύσεις για μια βιώσιμη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγγετριά μας είναι η κυρία Αντέα Μακιντάιερ. Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σπουδαίο γιατί αφορά την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της γεωργίας, τη γεωργία ακριβίας, την επιλεκτική κτηνοτροφία, την ε, προστασία των φυτών, γενετικές πτυχές, ε, γενετική μηχανική, αλλά και θέματα χρηματοδότησης ε, και σωστής αξιοποίησης των πόρων για την πρόθεση της καινοτομίας. Οπότε είναι ένα θέμα που περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Θα δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας για να μας κάνει μια εισαγωγή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ που αναβάλλατε το θέμα, ώστε να προλάβω να φτάσω και να σας κάνω την παρουσίαση. Το σημείο αφετηρίας ε, για την ε, έκθεσή μου είναι διπλό. Είναι η βιωσιμότητα και η παραγωγικότητα. Οι τεχνολογίες γεωργίας έχουν ε, τη δυνατότητα να κάνουν και πιο παραγωγική τη γεωργία, αλλά και πιο βιώσιμη, πιο αηφόρα. Πολλοί γεωργοί αντιμετωπίζουν τη τεχνολογία, δηλαδή τη γενετική, τη μηχανική, αλλά και τη ψηφιακή τεχνολογία ως το μόνο ρεαλιστικό τρόπο για να αντιμετωπίσουν ε, τις ε, περιβαλλοντικές προκλήσεις και την πρόκληση εξασφάλισης ε, των τροφίμων. Αλλά είναι σημαντικές και οι μη τεχνολογικές λύσεις για την εξασφάλιση της βιώσιμης γεωργίας. Για παράδειγμα, οδηγία για την βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων. Αναγνωρίζουμε επίσης τον κεντρικό ρόλο που έχει μια ολοκληρωμένη διαχείριση στα θέματα αυτά. Βέβαια, η χρήση τη τεχνολογία είναι ένα σημαντικό τμήμα τη λύση, χωρί να υποτιμούμε και τι άλλε πτυχέ, και επίση ζωτικό εργαλείο για να βοηθήσουμε του Ευρωπαίου γεωργού να προσαρμοστούν στι αρχέ τη ολοκληρωμένη διαχείριση ε, των φυτοφαρμάκων. Και εδώ έχουμε ιδιαίτερα τις τεχνικές ε, γεωργίας ακριβίας και για, τις, ε, και για τη γεωργία και για την κτηνοτροφία. Γιατί η γεωργία ακριβίας μπορεί να μειώσει τη χρήση των φυτοφαρμάκων, να μειώσει τη χρήση του ύδατος και να μειώσει και τη χρήση των λιπασμάτων. Ενώ θα βελτιώνει τη γονιμότητα των ε, εδαφών και βελτιστοποιεί τις εισοδηγές. Βέβαια το υψηλό κόστος αυτών των τεχνολογιών και η δυσκολία προσαρμογής των τεχνολογιών αυτών σε μικρές ε, γεωρικές εκτάσεις ε, με ακανόνιστες συνθήκες ε, είναι υψηλές. Μάλιστα δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών γεωργίας ακριβίας. Θεωρούμε ότι κυμαίνονται μεταξύ του 3 και του 8% τα ποσοστά χρήσης αυτών των τεχνολογιών. Ε, η έκθεσή μου δίνει έμφαση στον κεντρικό ρόλο που έχουν οι γεωργοί. Και ενώ οι γεωργικές τεχνολογίες αναπτύσσονται, δεν είναι όλες ικανές να ανταποκριθούν στις ανάγκες των γεωργών. Είτε γιατί δεν έχουν βελτιστιοποιηθεί ακόμα οι τεχνολογίες, είτε γιατί ε, απαιτούν μια ένταση κεφαλαίου. Οι γεωργοί όμως είναι οι τελικοί χρήστες αυτών των τεχνολογιών. Και οι γεωργοί θα πρέπει να εμπλέκονται την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών. Οπότε η ανάπτυξη των τεχνολογιών, των γεωργικών τεχνολογιών, θα πρέπει να αξιοποιεί και την πείρα των γεωργών. Οι γεωργοί θα πρέπει να αναμειγνύονται στην αλυσίδα της ανάπτυξης αυτών των γεωργικών τεχνολογιών και όταν ε, κάποιο γεωργό αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη πρόκληση, θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στην επιστήμη, στους επιστήμονες και να χρησιμοποιεί τη βασική έρευνα για να βρει λύση στα προβλήματά του. Επίση, ε, τα πλεονεκτήματα των καινοτόμων τεχνολογιών δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε ένα μόνο είδο γεωργική πρακτική οι τεχνολογίε θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα είδη γεωργία. Είτε είναι συμβατική αυτή η γεωργία, είτε βιολογική, είτε γεωργία, είτε κτηνοτροφία, μικρή ή μεγάλη κλίμακα. Θα πρέπει τα πλεονεκτήματα τη καινοτομία και τη τεχνολογική ανάπτυξη να είναι προσιτά σε όλου του γεωργού και κτηνοτρόφου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμω πολλά προσκόμματα. Πέραν των περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Γεωργία, οι επενδύσει στην έρευνα έχουν μειωθεί δυστυχώ ε, τα τελευταία 30 χρόνια παντού στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα η ικανότητα να ε, καλλιεργούμε περισσότερο ε, περισσότερα τρόφιμα έχει μειωθεί. Οπότε η παραγωγικότητα σε τρόφιμα δεν μπορεί να ενισχυθεί βιώσιμα χωρίς μόνιμες επενδύσεις στην βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα και η ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας αλλά και της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας δεν περιορίζεται στην οικονομία μόνο. Με 850 περίπου εκατομμύρια στον κόσμο να, να υποφέρουν από χρόνια υποσυτισμό, οι περισσότεροι μάλιστα διαβιούν στις αναπτυσσόμενες χώρες, δημιουργείται η ηθική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βελτιώσει την ιδιωτική της παραγωγή και να την αυξήσει με βιώσιμο όμως και υφόρο τρόπο. Οι πρόσφατες επενδύσεις σε κοινέ χρηματοδοτικές προτεραιότητες των κρατών μελών και των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα ρίνονται και χαίρομαι που ε, περιλήφθηκε στην πρόσφατη, στο πρόσφατο έγγραφο εργασίας για τον ορίζοντα 2020 και η γεωργία ακριβίας. Βέβαια, η εφαρμοστικότητα της τεχνολογίας θα κρίνει κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί αυτή από του Γιώργους. Γι' αυτό και ε, παραλαμβάνω, οι Γιώργοι θα πρέπει να αναμειγνύονται ενεργά στα σχέδια αυτά. Η έκθεσή μου αναφέρεται ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο ε, μνημόνιο Συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανάπτυξη τη υπαίθρου και τη Γεωργία για το 2020. Και μάλιστα η προστιθέμενη εξή αυτών των εργαλείων ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μόχλευση που δημιουργούν και τις εγγυήσεις που δίνουν για τα δάνεια, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Και αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση των επενδυτικών αναγκών των γεωργών και του κινδύνου σε ό,τι αφορά την τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Θα πρέπει φυσικά στα νέα προγράμματα ανάπτυξη πέστρων να συμπεριληφθούν και οι πρακτικέ αυτέ. Έχουμε πολλέ επενδύσει νέε και στα κράτη-μέλη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, η Βρετανική κυβέρνηση επενδύει σε μια νέα στρατηγική, Agritech, προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο να ε, πρωτοστατήσει σε ε, γεωργική καινοτομία και βιωσιμότητα. 70 ε, εκατομμύρια λίρες θερίνες χρησιμοποιούνται σε καταλήτες Agritech προκειμένου να επιταχυνθεί η εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της γερικής έρευνας. γιατί επίσης 90 εκατομμύρια λίρες τερλίνες στόχο έχουν ε, την ε, ε, χρήση της καινοτομίας στα θέματα αυτά προκειμένου να προσελκυστούν οι, κατάλληλοι, ε, οι κατάλληλες δεξιότητες και να προσελκυστούν κατάλληλα πρόσωπα και εμπειρογνωμοσύνη στον κλάδο. Οι ερευνητικέ ικανότητε που περνούνται για την υποστήριξη του τομέα μεταβάλλονται με ταχύ ρυθμούς και υπάρχει αυτή τη στιγμή πραγματικό κίνδυνο αύξηση των ελλείψεων σε ανώτερε δεξιότητε στην αγρονομία και στην πετοπαθολογία, καθώ πολλοί από του έμπειρου επαγγελματίε αυτού του εξειδικευμένου τομεί πλησιάζουν στη δεξιοδότηση. Σε μεγάλο μέρο τη Ευρώπη, τα κέντρα εκπαίδευση, κατάρτιση και καινοτομία έχουν υποβαθμιστεί και χρειάζονται αναζωογόνηση ιδιαίτερα στον αναδυόμενο τομέα της γεωρική μηχανικής. Εν συντομία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να κάνουν το γεωργικό τομέα της Ευρώπης πιο ελκυστικό για τους νέους ερχόμενους, είτε στη γεωργία, είτε στην έρευνα, είτε στην ανάπτυξη τεχνολογιών. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου που θα είναι πιο φιλικό προς τις επενδύσεις και ε, να φροντίζουμε ότι η κοινοτική νομοθεσία δεν δημιουργεί τροχοπαίδηση στη καινοτομία είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το νέο μηχανισμό επιστημονικής ε, παροχή συμβουλών για να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε επιστημονικά κριτήρια και να εξασφαλιστεί ε, η ισορροπία μεταξύ του ωφέλους και των κινδύνων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δημιουργία νέων προϊόντων προστασία ε, των φυτών και μία ολοκληρωμένη διαχείριση των φυτοφαρμάκων. Τέλος, η έκθεσή μου αναφέρει ότι η απώλεια βιοπικιλότητα του τελευταίο αιώνα υποβαθμίζει και υπονομεύει τις ευρωπαϊκές πολιτικές για μια βιώσιμη γεωργία και τονίζει την ανάγκη ενισχυμένου διάλογου, διαλόγου μεταξύ γενετικών τραπεζών και τελικών χρηστών, ώστε να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και να στηρίξουμε μια βιώσιμη παραγωγή τροφίμων σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι οι μακροπρόθεσμε προκλήσει τη βιώσιμη γεωργία πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια κοινή προσέγγιση τη Επιτροπή και των κρατών μελών για να εξασφαλιστεί η στήριξη τη τεχνολογική καινοτομία και περιμένω με ανυπομονησία τα σχόλια των συναδέλφων για την έκθεση καθώς και τις τροπολογίες τους στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματός μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολλοί συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ καθένας. Η ε, κυρία Μόλι Σκοτ Κάτο είναι η πρώτη. Ένα λεπτό παρακαλώ όμω. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εκπροσωπώντα την ομάδα των Πρασίνων, ξέρετε ότι ε, είμαστε υπέρ μια συγκεκριμένη τεχνολογία και είμαστε και υπέρ τη καινοτομία. Είναι το πιο σημαντικό όμω να έχουμε την απαραίτητη τεχνολογία. Μια τεχνολογία δηλαδή που θα συνάδει με τη φύση. Νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να πετύχουμε αν λειτουργήσουμε σε αρμονία με τα οικοσυστήματα και δυστυχώς αυτό δεν το βλέπουμε καθόλου σαν ιδέα στην έκθεση της κυρίας Μάκεντάιρ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα να μπορεί δηλαδή το έδαφος να απορροφά τόσο το νερό όσο και τον άνθρακα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά πρέπει και το έδαφος αυτό να είναι βιώσιμο, να ζει, να είναι γόνιμο, προκειμένου να έχουμε πραγματικά και μια βιώσιμη γεωργία. Και νομίζω ότι τα προβλήματα τα οποία ανέφερε η κυρία Μακιντάιερ έχουν να κάνουν πραγματικά με την ποιότητα του εδάφους και το γεγονός ότι δεν σεβόμαστε αρκετά το περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και αυτό ενταχθεί ιδέα. Η κυκλική οικονομία επίσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν έχουμε ένα υγιές οικοσύστημα. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε πόρους, έχουμε καλύτερο έδαφος και καλύτερη ανθεκτικότητα. Μπορούν οι Γεώργοι εδώ πέρα να επιφέρουν πολύ θετικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, αλλά όχι ακολουθώντα τα όσα λέγονται στην έκθεση αυτή, όσον αφορά τι νέες τεχνικές αναπαραγωγής. Μας προσκαλούν αυτές μια κάποια ανησυχία. Δεν θέλουμε τέτοιες νέες τεχνικές και δεν θέλουμε να χρησιμοποιείτε ούτε καν το MBT ως νέο αρχικό, γιατί έχουμε ήδη ένα αρχικό το GMO ουσιαστικά τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και ξέρετε ότι ήδη στην οδηγία για τα βιοτεχνολογικά προϊόντα έχουμε ήδη έναν, μια μνήμα στα προϊόντα αυτά. Και ξέρετε ότι επίσης η ΕΦΣΑ έχει αναφερθεί στον τρόπο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε μία διαφορετική προσέγγιση. Είπατε εσείς ότι αναφερθήκατε σε μία έρευνα η οποία συγκρίνει το πέμπτο και το έβδομο πρόγραμμα έρευνας και τη χρηματοδότηση της καινοτομίας. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπήρχε μια πολύ σημαντική μείωση των αρχικών ποσών που δόθηκαν, ενώ υπήρχε αύξηση στην έρευνα η οποία δόθηκε σε άλλου τομεί. Συγγνώμη επίση για τον αν μακρηγόρησα. Επαλαμβάνω το βασικό σημείο της παρεμβασίσμου. μου, είναι πολύ σημαντικό να λειτουργήσουμε σε αρμονία με τη φύση. Όχι μόνο ξεπεράσετε το χρόνο σας, αλλά ξεπεράσετε διπλάσιο από το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας. Ελπίζω να μην σας μιμηθούν οι άλλοι συνάδελφοι. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ε, ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Προσπαθώ ένα-δύο ζητήματα να εκθέσω. Στο σημείο ε γίνεται λόγος για την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων. που χρησιμοποιούνται περίπου για που για την Παρασκευή του χρησιμοποιείται περίπου το 5% τη ενέργεια από ορυκτά καύσιμα που καταναλώνεται από τα αισθήματα ιεροπή παραγωγή. Ε, η αεροβική επίση πέψη ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε. Μπορούμε να, σώσουμε, να λύσουμε πολλά προβλήματα. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα και να δημιουργούμε ενέργεια. Αυτό σημαίνει αηφορία. Στα κοινωνικά μέσα, στο marketing μπορούμε να έχουμε δυνατότητες για μικρούς παραγωγούς, μικρές εκμεταλλεύσεις να διαθέσουν ταχύτατα τα προϊόντα τους. Μπορεί κανείς να το κάνει και, με... και μέσα στο χώρο της πολιτικής. Εγώ το δικό μου το περιορισμένο μικρό προϊόν που δεν είμαι μεγάλο παραγωγός πολιτικής, το διαθέτω γρήγορα χάρη στο η τεχνολογία. Το ίδιο μπορεί και ο Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό με το Twitter κτλ. Να κοιτεί ε, ο άνθρωπος επίσης, ο πολίτης, να αγοράζει τον τόπιο προϊόν. Ο τουρίστας να αναζητεί τον τόπιο προϊόν. Χάρη στα ε, social media, Instagram, Twitter, ό,τι θέλετε. Αλλά μπορεί. Ευχαριστώ κυρία Γιλέρα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μακιντάιρ για το σχέδιο έκθεσής της. Πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση και σε πολλά σημεία συμφωνώ. Διαφωνώ με κάποια σημεία, αλλά με πολλά συμφωνώ και πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να έχουμε ειδική έκθεση της Επιτροπής μας που θα μιλά για την ανάγκη, την αναγκαιότητα της ε, τεχνολογικής καινοτομίας. Θα πρέπει να επενδύσουμε και να δώσουμε έμφαση στην ε, τεχνολογική καινοτομία για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα της γεωργίας. Χαίρομαι που το πραγματευόμαστε αυτό σε μια έκθεση. Και φυσικά να μην ξεχνάμε και τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο που μας δεσμεύει. Και αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου στο όνομα της βιωσιμότητας να μένουμε πίσω σε ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα θα πρέπει πολύ σοβαρά να ασχοληθούμε και να αναγνωρίσουμε την ανάγκη της τεχνολογικής καινοτομία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, η ανάγκη να αναθεωρηθεί το κανονιστικό πλαίσιο των φυτοφαρμακευτικών προϊόντων. Μόλις έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό τριμερής διάλογο για ένα τέτοιο θέμα και πιστεύω ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο και εκεί. Δυστυχώς εξάντλησα το λεπτό μου και δεν μπορώ να επεκταθώ σε άλλα σχόλια που επίση είναι σημαντικά. Αλλά συνοψίζοντας, να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον που λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτό το θέμα της ανάγκης της ε, ε, τεχνολογικής καινοτομίας και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στη βιωσιμότητα ξεχνώντας ε, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα. Κύριος Χαγουσλήμ, Πρόεδρε, με ξαφνιάζει λίγο το ότι συζητούμε ένα ζήτημα το οποίο είναι η δεύτερη φορά που το βλέπουμε μπροστά μας. Γιατί να μην αφιερώσουμε την εργατικότητά μας σε κάτι άλλο. Εμείς, Πρόεδρε, είχαμε ζητήσει κάποια άλλα θέματα που όμως δεν δεχθήκατε να μπουν στην ημερησία διάταξη, το υπενθυμίζω αυτό. Και βλέπουμε εδώ ότι κάποιοι θεωρούν πως η τεχνολογία μπορεί να τους λύσει όλα τα προβλήματα. Στο σχολείο όταν πήγαινα εγώ μου λέγανε «Α, ολοκληρωμένη γεωργική παραγωγή» αλλά κανείς δεν με εξηγούσε γιατί με την ολοκληρωμένη γεωργική παραγωγή όλο και περισσότερα ήταν τα, προς τα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούσαμε. Δεν είναι η τεχνολογία δηλαδή το πρόβλημα. Γιατί να μην διαθέσουμε περισσότερα κονδύλια για έρευνα στην βιολογική γεωργία που έχει λύσει πολλά προβλήματα μέχρι τώρα χωρίς τέτοια χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει δηλαδή στην απεικόνηση της υποστήριξης της έρευνας κάτι το οποίο να δείχνει πως υποστηρίχθηκε η βιολογική παραγωγή. Γιατί, γιατί η μεγάλη βιομηχανή παραγωγή είναι αυτή η οποία απομυζά τα κέρδη. Ευχαριστώ κυρία Ράς Γκαρσία. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την προσπάθεια που κάνει ε, και την αναγνώριση της σημασίας ε, των τεχνολογικών επιτευγμάτων για τη βιώσιμη γεωργία. Εγώ θα επικεντρωθώ στα φυτοφάρμακα, στα προϊόντα φυτοπροστασίας. Θα σας υποβάλω και τροπολογίες για το θέμα αυτό, γιατί θα ήθελα να επικαλεστώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάποιες μικρότερες καλλιέργειες, για τις οποίες επιβάλλαμε μόνοι μας απαγορεύσεις για ουσίες που προηγουμένως επιτρεπόταν και που έτσι στερούμε από τους γεωργούς τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν κάποιες ασθένειες των φυτών. Πρόκειται για μικρέ καλλιέργειε ίσονο που δεν είναι ελκυστικέ ακριβώ επειδή δεν έχουν μεγάλο κέρδο και τι έχουν εγκαταλείψει στη μοίρα του η επιστήμη και η τεχνολογική ανάπτυξη. Για να μην επαναληφθούν οι κίνδυνοι του παρελθόντο με οικειοθελεί απαγορεύσει που επιβάλαμε το 2005, ελπίζοντα το 2015 θα είχαμε την απαραίτητη επιστημονική έρευνα, προσοχή να μην την πατήσουμε και δεύτερη φορά και να αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον αντίστοιχα προβλήματα. Ο κύριο Σάντο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα με κάθε σεβασμό να πω ότι είμαι ο σκιώδης ηγητής των σοσιαλιστών ε, ε, για την έκθεση αυτή και δεν μου αρκεί ένα μόνο λεπτό και το λέω αυτό με κάθε σεβασμό κύριε Πρόεδρε. Έφυγα από άλλη συνεδρίαση, ήρθα εδώ, περίμενα τόση ώρα υπομονετικά ε, και ως και ο δεν πρόκειται να μιλήσω μόνο για ένα λεπτό, προτιμώ να μιλήσω καθόλου. Το λέω αυτό με κάθε σεβασμό, αλλά είναι απαράδεκτο να δίνουμε τόσο λίγο χρόνο για του και ηγητέ. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να μιλήσω καθόλου. Σα ευχαριστώ, αλλά έχουμε τόσο μακροσκελή κατάλογο αγόριτών. δεν προλαβαίνουμε περισσότερο χρόνο. Κύριο Σουλαζό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην έκθεση λοιπόν αυτή έχουμε την ίδια προσέγγιση με αυτή που έχουμε την έκθεση του κ. Γιάννη Τενάν, την οποία αντιμετωπίσαμε τον Ιανουάριο το ότι η κοινή γεωργική πολιτική αποτέλεσε αποτυχία δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κατακτήσουμε τι εξωτερικέ αγορές και να κάνουμε όλο και περισσότερες εξαγωγές. Βλέπω ότι υπάρχουν πολύ καλές προθέσεις, αλλά ουσιαστικά θέλετε να δημιουργήσετε εδώ πέρα ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι υπέρ τη βιομηχανία, απελευθερώνοντα ακόμα περισσότερο τι αγορέ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει την εργασία των γεωργών, δεν θα πρέπει, όπω είπα και στι 11 Ιανουαρίου, αυτό να αποτελέσει πρόσχημα για να μειωθεί ο ρυθμό των γεωργών και να αυξηθεί η συγκέντρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αν η έρευνα πρέπει να υποστηριχθεί, τότε θα πρέπει να εξυπηρετεί πραγματικά του γεωργού και όχι τη μεγάλη βιομηχανία, η οποία δεν τρέφεται τέτοια συμφέροντα και νομίζω ότι θα πρέπει μεγάλη αυτή η βιομηχανία να τεθεί υπό έλεγχο. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω με ποιο τρόπο μπορεί να εξασφαλίσετε ότι το σχέδιο σα αυτό δεν θα στρέφεται κατά των γεωργών, οι οποίοι εξαρτώνται πάρα πολύ από του μεγάλου βιομηχάνου, καθώ επίση και από του αρμόδιου στο χρηματοοικονομικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σουραπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, άλλε βουλέ ανθρώπων και άλλο Θεός και Λέβη. Γιατί εξετάζουμε τα στοιχεία και δημιουργούμε την ψευδέστηση ότι τα στοιχεία είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Πολλά έχουν γίνει ήδη και δεν θα πρέπει να θέτουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Πολλά κρατημέλη έχουν αποφασίσει να κλείσουν την πόρτα στους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Φαίνεται όμως ότι τώρα διαλέγουμε διαφορετικές κατευθύνσεις. Και δεν λέμε τίποτα πια για την βιολογική γεωργία ή τη βιώσιμη γεωργία. Μιλούμε για μη επικίνδυνα φυτοφάρμακα. Τι εννοούμε όμως. Πολλά ερωτήματα ανακύπτουν. Αλλά επαναλαμβάνω θα πρέπει να σκάβουμε μόνοι μας το λάκκο μας και να υπονομεύουμε το έργο που έχουμε ήδη κάνει. Ευχαριστώ, κύριε Σάγκνιο. Well, Κύριε Κάρφη, φαντάζομαι ότι θα σα ε, χαροποιήσει το γεγονός ότι υποστηρίζω τα σχόλιά σας σε σχέση με τις ειδωτικές μονάδες παραγωγής. Βεβαίω και η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγεί σε στασιμότητα την γεωργική παραγωγή. Είναι ξεκάθαρο αυτό με τους κανόνες που επιβάλλονται. Όλο και λιγότερα θα είναι τα ενεργά συστατικά που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τα φυτοφάρμακα. Θα αναπτυχθεί περισσότερη ανθεκτικότητα και μάλιστα εξάγουμε για αυτό το χειρότερο την αριστεία την επιστημονική σε άλλες χώρες για να εισαγάγουμε προϊόντα για να εισαγάγουμε αγιοργικά προϊόντα τα οποία έχουν τύχη υπεξεργασία σε άλλες χώρες με τα φυτοφάρμακα τα οποία στην Ευρώπη απαγορεύουμε. Παλαβομάρα δηλαδή. Όπως και να έχει. Ο παραγωγό ξέρει πολύ καλά να προστατευτεί, δεν τον κοροϊδεύουν οι μεγάλες εταιρείες, αν τον κοροϊδέψουν την πρώτη χρονιά, ναι, δύο δεύτερη χρονιά, ναι, αλλά όχι και την τρίτη, γιατί θα προστατεύσει τα συμφέροντά του και έτσι μπορεί να, ε, και έτσι πρέπει να τους βοηθήσουμε να δοκιμάζουν νέες ιδέες συμπεριλαμβανομένων και τη βιολογική καλλιέργειας. Ο κύριο Αντρίε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάκιντάιρ για την έκθεση. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις ε, η συγγήτρια επικεντρώνεται στην τεχνολογία, χωρίς ωστόσο να μας λέει σε τι τύπο γεωργίας ή σε ποιο μοντέλο γεωργικό σκοπεύει να προαγάγει τη χρήση της τεχνολογίας. Νομίζω ότι η τεχνολογία θα πρέπει να υπηρετεί με τις διαδικασίες της τη γεωργική παραγωγή για περισσότερη αηφορία. Και πρέπει να στραφούμε προς νέα μοντέλα πιο αηφόρου γεωργικής παραγωγής με την ιδέα της αγροοικολογίας, αγροοικολογίας. Δεν μπορούμε να μένουμε δέσμοι της θεώρησης και των προτύπων μιας βιομηχανικής μάλλον γεωργικής παραγωγής γιατί αναγκαζόμαστε την τεχνολογία να την προσαρμόσουμε σε αυτό το μοντέλο και έτσι δεν βοηθάει η τεχνολογία στην αλλαγή μοντέλου όπως είναι το ζητούμενο τώρα. Μιούλερ. Σύντομα, νομίζω ότι η καλλιέργεια των εδαφών μας με σεβασμό και οικονομική χρήση των πόρων συμπεριλαμβανομένων των υδάτων είναι πάρα πολύ σημαντική. Μια γεωργία με ακριβή και φιδωλή χρήση των πόρων είναι πάρα πολύ σημαντική και βέβαια νομίζω ότι θα έχει και μεγαλύτερη αποδοχή από τους πολίτες. Κυρία Μάκιντάιρ, διατυπώσατε πράγματι έκθεση αντίστοιχη με αυτή του συναδέλφου Γιάννη Κούτεμα. Για μένα σημαντικό θα ήταν να προβείτε σε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί του, έτσι ώστε να καθοδηγήσετε τα κείμενά σας προς την ίδια κατεύθυνση. Άλλωστε έχει και η Επιτροπή μας μια επίσκεψη στις κάτω χώρες, στο Βάγκενιγκεν. Και ίσως θα ήταν σκόπιμο οι, οι να συντονίσουν τις προσπαθίες τους για να μην επαναλαμβάνουν τα λόγια ο ένας του άλλου. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Μαγκίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την εισηγητριά μας. Πρέπει να σας πω ότι το επιστημονικό πάνελ ΣΤΟΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάνει αυτή τη στιγμή μια έρευνα όσον αφορά την γεωργία ακριβίας. Επομένω θα μπορούσαμε να έχουμε και από εκεί κάποια στοιχεία. Αναφέρατε επίση την έρευνα. Πολλά κράτη-μέλη έχουν μειώσει τη, τη χρηματοδότησή του προ την δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Επίση, η μεταφορά γνώσεων. Ξέρετε ότι πολλά κράτη-μέλη όπω και το Μένο Βασίλειο έχουν μειώσει τελικά, έχουν αναδιπλωθεί ...την μεταφορά αυτή γνώσεων προς τους γεωργούς. Οι γεωργοί πραγματικά θέλουν να έχουν περισσότερη γνώση, περισσότερη επιγνωμοσύνη. Πρέπει να υπάρχει όμως και το απαραίτητο σύστημα που να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Από ό,τι φαίνεται μπορεί να υπάρχει μια αντιπαράθεση ανάμεσα στις διαφορετικές προσεγγίσεις. Αναφέρεστε όμως εδώ πέρα σε τεχνολογικές λύσεις για μια βιώσιμη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι εδώ πέρα καλύπτεται και η εντατική γεωργία και η συμβατική και η βιολογική. Νομίζω ότι και οι τρεις μορφές γεωργίας θα πρέπει να καλύπτονται από την έκθεση αυτή. Η γεωργία χρειάζεται νέες ιδέες προκειμένου να εξελίσσεται και να είναι πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Ο Μπράνεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά άκουσα ότι η κυρία Μακιντάιρ αναφέρθηκε στο ότι μπορούμε να έχουμε και μη τεχνολογικές λύσεις στη γεωργία. Και έχοντας αυτό κατά νου, εγώ σκέφτομαι κατευθείαν τον αγροδασοκομικό τομέα. Αυτή την Παρασκευή θα πάω στην, στο αγρόκτημα του Στίβεν Μπρίξης. 125 εκτάρια είναι αν θέλετε η μεγαλύτερη αγροδασοκομική εκμετάλλευση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και με ιδιαίτερη χαρά να δώσω περισσότερες πληροφορίες στην Άνθεα μετά την επίσκεψη αυτή και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο και για τον πραγματικό ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία. Όντως, ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τεχνολογία θα πρέπει να εξυπηρετεί τη γεωργία και όχι η γεωργία να εξυπηρετεί την τεχνολογία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ζήτησε επίτηδες το λόγο άργα περιμένοντας μήπως έρθει ο σχέδιος συγκητής μας ε, πιο νωρίς. Ε, πάντως ευχαριστώ την κυρία Μάκιντσα για την πολύ θετική συνεργασία. Η γεωργία ακριβίας είναι εκ των όνου κάνε φόρο, όρος για την αηφορία στη γεωργία. Η γεωργία πρέπει να γίνει πιο ελκυστική για το εργατικό δυναμικό. Πρέπει να ωφεληθεί και ο μικροπαραγωγός στην απομακρυσμένη περιοχή της Υπέθρου. Η διατάξει Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να ε, παρεμποδίσουν την καινοτομία, άρα πρέπει να είναι πιο περιορισμένη η γραφειοκρατία. Η γενετική πολυμορφία επίσης είναι απαραίτητη. Στην γεωργία ακρίβειας πρέπει να είμαστε σε θέση να συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση της αηφορίας. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Βερολίνο είδαμε μεγάλες επιχειρήσεις στις εκθέσεις, αλλά νομίζω ότι τώρα πρέπει να δούμε και μικρές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην καινοτομία. Ευχαριστώ κύριο Γιάουρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ό,τι και να πούμε για τη σημασία της τεχνολογίας στη γεωργία, ε, πάλι δεν αρκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντική προφανώς. Είναι απαραίτητο, νομίζω, να και το αναφέρουν και οι συνάδελφοι, να μην γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ μικρού και μεγάλου. Δεν μπορούμε να κάνουμε ε, διαφοροποίηση μεταξύ εντατικής ή οικολογικής γεωργίας. Η γεωργία εν όλο έχει ανάγκη και απέτηση ε, από την υποστήριξη της τεχνολογίας και της επιστήμης. Άλλωστε, την παράθεση μεταξύ βιομηχανία και γεωργίας δεν βλέπω στην υπόθεση αυτή. Πρέπει να είναι συμπληρωματικές οι δράσει. Η τεχνολογία, η τεχνολογική εξέλιξη βιομηχανία είναι θετική και για τη γεωργία και νομίζω ότι αυτό το έναυσμα που δίνει η συγκεντρία είναι πολύ θετικό και πρέπει να το προωθήσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Εξαντλήσαμε το κατάλογο των ομιλητών. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Σάντος, στο μέλλον θα δίνουμε στους και ε, που ασχολούνται με συγκεκριμένο θέμα και που ουσιαστικά τις ομάδες του περισσότερο χρόνο. Έχετε δίκιο ότι κανονικά θα έπρεπε να έχει αφιερωθεί περισσότερος χρόνος για τους και ε, σας ζητώ συγγνώμη που δεν σας ε, έδωσε περισσότερο χρόνο. Στο μέλλον θα φροντίσουμε να το εξασφαλίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την προθυμία να λάβετε υπόψη το σχόλιο μου. Ωραία, ευχαριστώ. Ο κύριος Δημήτρου έχει το λόγο. Θα μπορούσε πραγματικό πολύ συμπυκνωμένα να κάνει κάποιο σχολιασμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την εισηγητρία για την ε, πρωτοβουλία που ανέλαβε να θέσει αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για τη γεωργία προς συζήτηση. Σημείωσε το σχόλιο και προσβλέπω την περαιτέρω συνέχιση των συζητήσεων. Ε, αναφέρονται σε πολύ συγκεκριμένε τεχνολογίε, ε, νέε τεχνολογίε αναπαραγωγή, ε, γεωργία ακριβία. Όλε οι τεχνικέ αυτέ είναι σημαντικέ και θα διδραματίσουν ρόλο στο να βοηθήσουν τον γεωργικό τομέα να αναπτύξει νέα προϊόντα, νέε υπηρεσίε και να ενισχύσουν την αγροτική οικονομία, δημιουργώντα θέσει απασχόληση. Η νέα πολιτική ανάπτυξη και η νέα στρατηγική το 2020 στηρίζουν την καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Αυτό αναφέρθηκε και εδώ. Η προσοχή που θα πρέπει να δώσουμε στην έρευνα και στο νέο ερευνητικό πρόγραμμα για τη βιολογική γεωργία. Ε, ο ορίζοντα 2020 και οι κοινωνικέ ε, προκλήσεις που επίση πραγματεύεται ε, υιοθετεί μια προοδευτική προσέγγιση και για τη γεωργία και μια σταδιακή αύξηση του προπολογισμού. Και μάλιστα αυτό προβλέπει και το πρόγραμμα εργασιών ε, για το 2016-2017. Να δώσουμε μεγαλύτερη ε, θέση και σημασία στη βιολογική γεωργία με περισσότερο προπολογισμό. Είναι σημαντικό να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ βιωσιμότητα και παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητα. Και ε, χαίρομαι για το θέμα αυτό που θέσατε στην έκθεση πρωτοβουλίας. Επίσης, δικαίωμα του Γεωργού να έχει πρόσβαση στα επιστημονικά πορίσματα και να έχει άμεση επαφή με τους επιστήμονε. Και μάλιστα προβλέπεται κάτι τέτοιο στην ευρωπαϊκή πολιτική, άμεση πρόσβαση των γεωργών στους επιστήμονες. Και μάλιστα 94 ε, προγράμματα αναπτυξιακά στηρίζουν τέτοιες δράσεις και περιμένουμε 3.200 πιλωτικά προγράμματα από τι 24 χώρε μέλη που έχουν προγραμματίσει αυτή τη δραστηριότητα. Και μάλιστα το σχέδιο έκθεση μιλά για την ανάπτυξη ενό ευρωπαϊκού κέντρου πρόθεση τη γεωργική καινοτομία. Ήδη έχουμε προβλέψει κάτι τέτοιο και μάλιστα με ελαστικό τρόπο και δημιουργία θεματικών δικτύων. Τα δίκτυα αυτά δημιουργούν πανευρωπαϊκά συστήματα δεδομένων για τέτοιες γνώσεις που μπορούν να, να χρησιμοποιηθούν άμεσα από όλους τους γεωργούς. Σε ό,τι αφορά την πολιτική ορίζοντα 2020, ε, ο Επίτροπος Χόγκαν θα, κάνει, διοργανώσει μια συνδιάσκεψη για τη γεωργική αυτή προσέγγιση και την καινοτομία στο τέλη της εβδομάδας. Και ε, εκεί θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του κλάδου, και φυσικά είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε περαιτέρω την ερευνητική μας πολιτική και στη γεωργία. Και σας διαβεβαιώ ότι πολλά από τα θέματα που σήξατε θα καλυφθούν και στη διάσκεψη που θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας. Θέλουμε κάποιες τεχνικές λύσεις για να προωθήσουμε μια βιώσιμη γεωργία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η συγκεκριά μας, η κυρία Μάκιντάιρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν το λόγο για να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι με βοηθάει πάρα πολύ αυτό και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία με όλους σας. Θα ήθελα απλώ να τονίσω κάποια ζητήματα τα οποία έθιξα πριν από λίγο στην αρχική μου παρέμβαση. Οι τεχνολογίε πρέπει να αναπτυχθούν για όλε τι μορφέ τη γεωργία. Τη συμβατική, τη βιολογική, μικρής, μεγάλης κλίμακας και τα λοιπά. Σαφώς δεν θα πρέπει η τεχνολογία να περιοριστεί σε μία μορφή γεωργίας. Προφανώς λοιπόν μπορούμε να έχουμε τεχνολογικές λύσεις για τη βιολογική για παράδειγμα γεωργία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να μην γίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα κάποιες από τις ρομποτικές λύσεις που έχω δει, κάποια ρομπότ τα οποία βγάζουν κάποια ζυζάνια, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στη βιολογική γεωργία. Θα ήθελα Επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Γκαρθία και προσβλέπω πραγματικά στις τροπολογίες σας για τις εξειδικευμένες καλλιέργειες και για την προστασία τους. Ξέρετε ότι στη δική μου την περιφέρεια υπάρχουν πολλές τέτοιες. Προσβλέπω πραγματικά στις τροπολογίες σας. Αναφερθήκατε επίσης, κυρία Μαγκίνες, στο πάνελ ΣΤΟΑ Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όντω να του συμπεριλάβουμε. Δεν υπάρχει λόγο να ξεκινάμε κάθε φορά από την αρχή. Α λάβουμε υπόψη μα τα πορίσματα τα οποία είναι σε θέση ήδη να μα δώσει η ΣΤΟΑ. Συμφωνώ επίση με τον Στιουαρτ Agnew ότι θα πρέπει προφανώ να αναφερθούμε σε όλου του καινοτόμου γεωργούς, να του περιλάβουμε στα προγράμματα αυτά και θα πρέπει επίση να δούμε τι γίνεται όντω και με τον τομέα τη δασοκομεία. Δώστε μου και γι' αυτό σα παρακαλώ περισσότερα στοιχεία και επίσης ε, για όσα δεν έχω συμπεριλάβει στην έκθεσή μου ή δεν μπορώ να καλύψω αυτή τη στιγμή σας διαβεβαιώ ότι έχω κρατήσει πολύ λεπτομερείς σημειώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ. Πραγματικά κρίμα που τα ρομπότ που ξεριζώνουν ζυζάνια δεν ε, χρησιμοποιούνταν και όταν εγώ ήμουν μικρός και ε, χρειαζόταν ως παιδάκι να πηγαίνω και με τα χέρια μου να ξεριζώνω τα ζυζάνια από τα χωράφια. Λοιπόν, διορία για την υποβολή τροπολογιών. 29 Ιανουαρίου στι 12 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Σα ευχαριστώ όλου για τη συζήτηση και περάμε στο σημείο 9, τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή των Άλπαιων. Συντάκτηρια γνωμοδότη είναι η κυρία Ουλρίκε Μίλλερ. Έχουμε την τέταρτη μακροπεριφερειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που αφορά την περιοχή των Άλπαιων αυτή τη φορά και παρόλο που έχουμε στρατηγική νέα, δεν έχουμε νέα και πρόσθετα κονδύλια. Ουσιαστικά προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνέργεια μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που προβλέπονται σε διάφορους μηχανισμούς. Δεν προβλέπονται νέα πρόσθετα κονδύλια. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα περιφερειακά προγράμματα, τα μακροπεριφερειακά προγράμματα και θα πρέπει να τα μελούμε. Θα μας τα πει όμως καλύτερα η συντάκτη της γνωμοδότησης, η κυρία Μίλλερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Θέλω καταρχάς να ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προετοιμασία μη στρατηγικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αλπικές ζώνες που έχει ετοιμάσει. Αυτή είναι η βάση της ανακοίνωσης. Την καλωσορίζω. Στην ε, αλπική περιοχή των, ε, της Ευρώπης έχουμε 7 κρατημέλη, 80 εκατομμύρια πολίτες, 48 περιφέρειες. Και ξέρουμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση η αλπική περιοχή. Είπατε και εσείς στην εισήγηση ότι δεν πρόκειται να δοθούν νέα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του υφισταμένου ε, νομικού πλαισίου θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, αλλά εγώ ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι σε ένα σκόπιμο, χάρη στο πρόγραμμα Interreg, που δρά και υπερσυνοριακά, να βρούμε λύσεις ε, και για την περιοχή των Άλπαιων, που θα καλύπτει έτσι και το χώρο της γεωργίας, με υπερσυνοριακά έργα που μπορούμε στοχευμένα να υποστηρίξουμε. Είναι γνωστή η αλπική ζώνη, την γνωρίζουμε και την αγαπάμε όλοι. Είναι αδιανόητο να συνεχίσει να υπάρχει αν δεν υπάρχει γεωργία με τις σκληρές αυτές τοπογραφικές και ε, κλιματολογικές συνθήκες και τις οικογένειες που ζουν εκεί δουλεύοντας σκληρά κάθε μέρα που συμβάλλουν τον τρόπο αυτό στη διαφύλαξη της παραδοσιακού τοπίου, των, ε, ενός υγιούς οικοσυστήματος και των παραδοσιακών τροφίμων. Είναι απαραίτητο να οριστούν τα ορόσημα για τη συνέχιση αυτών των δραστηριοτήτων ε, των γεωργικών και για το μέλλον, ώστε να δοθούν προοπτικές και για τους νέους. Σημαντικό κατά είναι να κάνουμε πολιτική συγκεκριμένα για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτήν την γεωγραφική ζώνη, για τις οικογένειες, για τους ε, κατοίκους των περιεχών αυτών. Μια συγκεκριμένη και κοινή δράση από τα κράτη-μέλη που... στα οποία και η αλπική ζώνη. Πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε γνωμοδότηση εκ μέρους της Γεωργικής για την Περιφερειακή Επιτροπή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ε, γεωργικές δομές ε, ε, που ανέρχονται σε ετηρίδε, πρέπει να διαφυλαχθούν. Έχουμε να κάνουμε με μορφές κτηνοτροφίας παραδοσιακές. Έχουμε να κάνουμε με ένομες τάξεις κρατών μελών και ευρωπαϊκή ευρωπαϊκές ρυθμίσεις ε, και νομοθεσία που πρέπει να συνδυάζονται. Πρέπει να έχουμε τη διασταυρούμενη συμμόρφωση για τις ε, εκμεταλλεύσεις στις περιοχές αυτές. Να, πρέπει να προστατέψουμε τα δάση και τα εδάφη, η αξιοποίηση δηλαδή και η εκμετάλλευση να γίνεται κατά λόγο ορθολογικό ώστε να διαφυλάσσεται και η βιοποικιλότητα και το τοπίο και η υδάτινοι πόρη. Η αηφορία στη χρήση των πόρων σημαίνει ταυτόχρονα και καλύτερη εξασφάλιση, μεγαλύτερη εξασφάλιση παραδοσιακών μορφών και πάνω απ' όλα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Ιδιαίτερα εγώ ενδιαφέρομαι για την προστασία των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, των μικρών οικογενειών, των οικογενειών που έχουν μικρές εκμεταλλεύσεις και βέβαια οι οδηγίες σχετικές με το ενδιέτημα, με την προστασία χλωρίδας και πανίδας, με την απαγόρευση των αζωτούχων λοιπασμάτων θα έχουν εδώ εφαρμογή. Οι κλιματικές αλλαγές σημαίνουν πολύ μεγάλες πολύ μεγάλους κινδύνους είτε από χιονοστιβάδες είτε από πλημμύρες ε, για τις ε, αλπικές ζώνες. Χρειάζεται πολιτική για τον άνθρωπο στις αλπικές ζώνες. Ε, ελκυστική δηλαδή, ελκυστικές συνθήκες διαβίωσης, ανταγωνιστικές συνθήκες διαβίωσης, δηλαδή και κινητικότητα και ψηφιακές υποδομές και προμήθεια ενέργειας, αλλά εν τέλει και βελτίωση κοινωνικών δομών και, και εξασφάλιση της χρήσης των γεωργικών γεών. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο στις προτάσεις μου. Ε, προσπαθούμε να στρέψουμε το βλέμμα και προς την εκπαίδευση, την έρευνα, την ανάπτυξη, γιατί έχουμε πολύ καλές, ε, καλούς συνδετικούς ε, ε, κρίκους στο χώρο της ε, υπαίθρου, της ανάπτυξης υπαίθρου στους, για τους τομείς αυτέ, αυτούς και μπορούμε να εξασφαλίσουμε δυνατότητες ε, και απασχόλησης που θα επιτρέπουν στο μέλλον στους νέους μας να παραμένουν στις περιοχές αυτές της υπαίθρου. Πολλές είναι οι προτάσεις, περιμένω βέβαια και τις προτάσεις των συναδέλφων και τις ενδεχόμενες προτάσεις για τροπολογίες, θα τις δεχτούμε με μεγάλη ευχαρίστηση, ώστε να έχουμε στο δυνατόν πιο καλή ε, έκθεση από πλευρά τη Επιτροπής, γνωμοδότηση από πλευρά τη επιτροπή Γεωργίας. Ευχαριστώ. Τέσσερις συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Άλλος κανείς? Όχι, οπότε 1,5 λεπτό καθένα. παρακαλώ. Κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ εδώ πέρα τον κύριο Ντόρφμαν, ο οποίο είναι ο σκιώδη ο οποίο δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ πέρα σήμερα. Επομένω, <laughs> μην πυροβολήσετε εμένα. Μιλάω εξ ονόματο του κυρίου Ντόρφμαν, όπω σα είπα. Οι μακροπεριφέρειε και σχετική στρατηγική έχουν ως στόχο να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τους υφιστάμενους σπόρους, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε διάφορα εδαφικά ζητήματα στα πλαίσια μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Η συγκεκριμένη αυτή στρατηγική για τις Άλπεις συνάδει με τη στρατηγική που έχουμε για το Δούναβι ή για τις Βαλτικές χώρες. Εν προκειμένου όμως η Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Ένωσης για την περιοχή των Άλπαιων θα επηρεάσει περίπου 80 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε 48 περιφέρειες, σε 7 χώρες εκ των οποίων 5 και είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Σλοβένια και δύο τρίτες χώρες, Λιχτεστάν και Ελβετία. Θεωρούμε λοιπόν ότι η μακροπεριφερειακή στρατηγική για τις Άλπεις θα πρέπει να συντονίσει τα, τους διαθέσιμους πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής, προκειμένου να εφαρμοστούν συγκεκριμένα προγράμματα στην περιοχή αυτή και να αντιμετωπιστούν προκλήσεις όπως προστασία του περιβάλλοντος, επενδύσεις στην καινοτομία, επενδύσεις στη γεωργία, τη δασοκομεία, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού. Θεωρούμε ότι ε, δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να δοθεί μια νέα χρηματοδότηση στα πλαίσια τη στρατηγική αυτή, αλλά θα πρέπει να συντονιστούν καλύτερα τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σουλαζό. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Πώς θα καταρτήσουμε μια κοινή στρατηγική για τόσο διαφορετικά, διαφορετικές περιφέρειες ε, με τόσο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι Γαλλικές Άλπεις ίσως είναι ένα εργαστήριο για τη μελλοντική γεωργία. Μικρές, ε, μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις ε, προσανατολίζονται στην τόπια αγορά με ισορροπημένη χρήση του εδάφους και με πρόσθετο ανοιχτού ε, τοπίου. Η εποχική απασχόληση είναι σταθερή. Το πρόβλημα είναι με τα εισοδημάτια, γιατί οι μικρές ε, εκμεταλλεύσεις έχουν ε, πολύ έθραυστα και ευάλωτα εισοδήματα και μάλιστα έχουν μειωθεί. Ε, κυρίως πλήττονται από μια προσπάθεια συγκέντρωση. Άλλο αρνητικό αποτέλεσμα είναι το, η επιδείνωση περιβαλλοντική. Και αν ε, έχουμε κάποιες ε, ε, ενισχύσεις που ενισχύουν την ελεξάρτηση, αυτό δεν θα είναι καλό, γιατί η αλπική οικονομία στρέφεται κυρίως σε μικρά κυκλώματα προσπαθούσε να καταπολεμήσει αυτή την συγκέντρωση και μάλιστα έχουμε πολλές α, ονομασίες προέλευσης ελεγχόμενης ή προϊόντα βιολογικής γεωργίας ή εμπορευματοποίηση σε πολύ μικρό κύκλωμα. Αυτό είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ελπικής οικονομίας. Πώς θα διαφυλάξετε τις ιδιαιτερότητες της ελπικής οικονομίας και τις τοπικές διεξόδους που αναζητεί, γιατί προσανατολίζεται κυρίως στις εγχώριες τοπικές αγορές. Ευχαριστώ. Κύριε Αγγιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η στρατηγική για την περιοχή των Άλπαιων. αλλά μας ε, δείχνει κάποιες προσπάθειες ε, συντονισμού και πολιτικής δράσης σε μια ορεινή περιοχή, γιατί η Άλπης είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Τώρα βλέπουμε τον οικονομικό τομέα και πώς ε, συνδυάζεται με τον τουριστικό ή με τον γεωργικό τομέα. Ταυτόχρονα γίνεται μια ανάλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η περιοχή αυτή των Άλπαιων, κυρίως ε, δυσκολίες μεταφοράς, ε, κάποιες κοινοφελείς υπηρεσίες, επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα ακόμη και βασικές στοιχειώδεις υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν να ευθετήσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την περιφέρεια αυτή και να συντονίσουμε την πολιτική μας δράση. Ε, Μερικέ φορέ δεν χρειαζόμαστε επιπλέον πόρου, αλλά καλύτερη αξιοποίηση των υφισταμένων πόρων. Γιατί ε, τα προβλήματα τη περιοχή των Άλτων είναι χαρακτηριστικά προβλήματα οποιασδήποτε ορεινή περιοχή, που είναι η εγκατάλειψη, απερίμωση, αν δεν έχουμε τι ε, επαρκείς υπηρεσίε και τη στήριξη στον τοπικό πληθυσμό, ώστε να παραμείνει στι ορεινέ περιοχέ. Η γεωργία, η ορεινή γεωργία, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν χρειαζόμαστε όμω μια κατακαιρματισμένη προσέγγιση, αλλά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τι ιδιάζουσε αυτέ ζώνε και τον τομέα τη γεωργία αυτέ. Και μάλιστα έχουμε 80 εκατομμύρια ανθρώπου που διαβίουν στην περιοχή των Άλπων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώ θα εφαρμόσουμε αυτή τη στρατηγική ώστε να μεταφέρουμε τι εμπειρίε τη και σε παρόμοιε ορεινέ περιοχέ στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριο Ντέ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την κυρία Μίλλερ για την έκθεση αυτή, την οποία υποστηρίζω ανεπιφύλακτα. Πρέπει ιδιαίτερα να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για τους ε, κτηνοτρόφους, για τους αγρότες στις ορεινές αυτές περιοχές, γιατί παραμένουν εκεί υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και πρέπει βέβαια να εκφράσουμε την ευχή να παραμείνουν εκεί. Βλέπουμε ότι όταν ε, εγκαταλείπει τις ε, ορεινές περιοχές ο αγρότης συχνά αλλοιώνεται προς το δυσμενέτερο και το περιβάλλον. Μπορούν, ξέρουν και θέλουν να διαφυλάσσουν ακόμα και για τον τουρίστα το περιβάλλον αυτό το αλπικό. Θα θυμηθώ την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, όπου ο κύριος Σόλος προσπαθούσε να μας πείσει ότι πρέπει μέσα σε τέσσερα εκτάρια να καλλιεργούνται στις αλπικές ζώνες πάνω από τρία διαφορετικά είδη οπόρων. Κάτι το αδύνατο. Φύση αδύνατο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ε, παραμένουν αυτοί οι παραγωγοί λοιπόν στις, οδικές, στις ορεινές ε, περιοχές Θέλω κλείνοντας ε, να πω ότι η ε, παραγωγή Φερρυπίν στο Βόρειο Τυρόλο έχουν μπορέσει να κρατήσουν μακριά από τις, ε, από τα χαμηλότερα, τις χαμηλότερες περιοχές και τον λύκο. Και αν σταματούσαν να δουλεύουν τις επιχειρήσεις τους, θα είχαμε τέτοια προβλήματα. Ο Διευθυντής τώρα, κ. Δημήτρη, εκ τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, όσο πιο λακωνικό είστε, τόσο περισσότερο θα το εκτιμήσουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η στρατηγική που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει ένα πλαίσιο για συλλογική δράση. Η ΚΑΠ εν όλο προσφέρει ευρύ φάσμα εργαλείων για την υποστήριξη των ε, αλπικών ζωνών. Αυτή η μακροστρατηγική έχει να κάνει με την καλύτερη ανάπτυξη των περιοχών, έχει νέα στοιχεία για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 για την κρηματοδότηση. Ή δείχνουν ότι όντως υπάρχουν πολλοί τομείς, φερρυπίν, επικοινωνίες, ε, επικοινωνιακές υποδομές που χρειάζονται υποστήριξη. Πέντε είναι τα κράτη-μέλη τα οποία καλύπτονται από την ε, αλπική ζώνη και έχουν αντίστοιχα διαπεριφερειακά προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο περιφέρειας ζητεί πρώτα από τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν τις εθνικές στρατηγικές και τις, σχέσεις, ε, και τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για να προχωρήσουν μετά στην υλοποίηση. Πρέπει τα προγράμματα για την ανάπτυξη πέθρου να προσαρμόζονται με μια οικολογική ε, λογική σε σχέση με διαφορές εδαφικές, ε, με τα χαρακτηριστικά. Η συνέπεια και η συνοχή έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τις ε, στρατηγικές με βάση και τα όσα υποστηρίζουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και πρέπει να υπάρξει ε, ανταπόκριση στα προγράμματα αυτά. Η ενίσχυση των στρατηγικών, η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ διαφόρων ε, μέσων χρηματοδότησης, το Περιφερειακό Ταμείο και άλλα έχουν βοηθήσει την ε, συνεργασία πέραν των συνόρων, καλύτερη συμπληρωματικότητα μεταξύ των ταμείων, ιδιαίτερα σημαντική για τομείς ευαίσθητους όπως οι υποδομές στην Ήπεθρο, η ευρυζωνικότητα, οι τοπικές υπηρεσίες. Η ανάπτυξη Πέθρου πρέπει να εστιάσει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της αρπικής περιοχής, επενδύσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταφορά μεταγνωσίας, υποστήριξη νέων γεωργών, γεωργικό, οικολογικά μέτρα, ομάδες παραγωγών, αλυσίδα παραγωγής, τοπικές αγορές και πολλά άλλα. Μεγάλη σημασία έχει βέβαια και η διασφάλιση ε, σταθερών πληρωμών με υποστήριξη του εισοδήματος των γεωργών στις περιοχές αυτές. Η ανάπτυξη μέσα από το πρόγραμμα Lidl σε υποπεριφερειακό επίπεδο μπορεί να συμβάλλει σε μια ισορροπημένη ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου στην αρπική ζώνη να ενισχύσουν τη συνοχή την εδαφική και την αηφορία Επίσης, μπορούν να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρων και να εξασφαλίσουν και καλύτερο συντονισμό και συμπληρωματικότητα σε σχέση με άλλα ταμεία. Στα σχέδια συνεργασίας για την υπαίθρο μεταξύ διαφόρων κρατών μελών ή και τρίτων ε, κρατών με διασυνοριακή συνεργασία μπορούμε να υποστηρίξουμε σχέδια που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ολυμπική Ζώνη. Περιμένω να συνεργαστούμε πολύ καλά με όλους εσάς για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σύντομα. Ε, σύντομα και ευχαριστώ πολύ. Πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες. Προσφέρω από σε καλή συνεργασία η μεταφορά γνώσεις μεταξύ των κρατών έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Μπορεί ο ένας δηλαδή να μάθει από τον άλλον. Ε, βέβαια δεν ξέρω πώς μπορούμε να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένα προγράμματα ή μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να στηρίξουμε στοχευμένα και μάλιστα μεταξύ ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών κρατών ε, ή ας πούμε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα στόχευαν σε συγκεκριμένε περιοχέ και προϊόντα συγκεκριμένων περιοχών, ενδεχομένω με ονομασία προελεύσεως. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Εγώ από τη δική μου την περιοχή μπορώ να πω ότι στο Αλγκόι έχουμε 600% ασφάλεια προμήθεια σε γάλα. Έχουμε μια πολύ καλή, καλά λειτουργούσα γεωργική οικονομία, μικρές δομές διάθεσης στην αγορά που λειτουργούν και μέσω του διαδικτύου, στέλνουν τα τυροκομικά προϊόντα Φερρυπίν και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ καλά στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις και 15 Μαρτίου θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε. Και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές ε, ανήκουν στην πολιτική συνοχή. Δεν θα πρέπει όμως να αυτή και τα συμφέροντα της γεωργίας. Γιατί η γεωργία, ιδιαίτερες ορεινές περιοχές, ε, γίνεται σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στη συζήτηση. Ευχαριστούμε την εισηγήτριά μας, συντάκτρια γνωμοδότηση ομάδα, Και περνάμε στο σημείο 10. Στην ανταλλαγή απόψε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Τζον Κλάρκ. Θα θυμάστε ότι στα τέλη ε, του προηγούμενου χρόνου είχαμε ε, κάποια ενημέρωση για την πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Αυτή τη φορά θα μας ενημερώσει ιδιαίτερα για το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων που για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ιδιαίτερη σημασία. Μια και δύσκολο είναι μερικές φορές να διεισδύσουμε στην παγκόσμια αγορά. Αυτό έχει δείξει και η διαπραγμάτευση του, της συμφωνίας TTIP. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευκαιρία ανταλλαγή απόψεων και δίνω το λόγο στον κύριο Κλάρκ. Well, thank, you very much, uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τζον Κλάρκ ονομάζομαι. Είμαι υπηρεσιακό αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Άγκρη και θα σα κάνω μία σύντομη παρουσίαση για τη διεθνή διάσταση των γεωγραφικών ενδείξεων, ένα ζήτημα το οποίο μα απασχολεί όλου, θεωρώ, στην αίθουσα αυτήν. Καταρχά, λοιπόν, θα πρέπει να θυμηθούμε λίγο τι είναι η γεωγραφική ένδειξη. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αναγνωρισμένη μορφή πνευματική ιδιοκτησία αντιστοιχεί ουσιαστικά στο copyright, στα δικαιώματα του δημιουργού ή σε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Πρόκειται για μια αγροτική, αν θέλετε, πνευματική διοκτησία. Πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο παράγεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή σύμφωνα με μια συγκεκριμένη μέθοδο παραγωγή ή σύμφωνα με μια συγκεκριμένη τεχνική και οδηγεί σε μια συγκεκριμένη ποιότητα, σε συγκεκριμένη φήμη για το προϊόν αυτόν, το οποίο συνδέεται με συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Και το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της γεωγραφικής ένδειξης είναι αυτή η αιτιώδη συνάφεια που υπάρχει ανάμεσα στο προϊόν, το όνομά του και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία παράγεται. Οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι πολύ σημαντικές από εμπορικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν είμαστε μόνο μεγαλύτερος εισαγωγός τροφίμων, γεωργικών προϊόντων, αλλά και ο μεγαλύτερος εξαγωγός τέτοιων προϊόντων και αυτό εν μέρη οφείλεται στις πολύ επιτυχείς μεταρρυθμίσεις της κοινή γεωργικής πολιτικής ή οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι έχουμε μια γεωργική πολιτική η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στην αγορά. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε τρόφιμα και προϊόντα τα οποία είναι περισσότερο από ποτέ τα αγωνιστικά στις διεθνείς αγορές. Έχουμε ένα εμπορικό ισοζύγιο πολύ σημαντικό της τάξης των 80 δισεκατομμύρων ευρώ σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και αυξήθηκε αυτό κατά 6%. Αυξήθηκαν οι εξαγωγές μας κατά 6% από πέρυσι και οι γεωγραφικές ενδείξεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό τμήμα των εξαγωγών αυτών. Όσον αφορά το εμπόριο σε προϊόντα που καλύπτονται από γεωγραφικές ενδείξεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η αξία των συνολικών προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων που εξάγαμε προς το εξωτερικό πέρυσι και παρά την απαγόρευση της Ρωσίας, το εμπάργο στη Ρωσία. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι οι γραφικές ενδείξεις συνδέονται με την πολύ μεγάλη ποιότητα που έχουν τα τρόφιμα και τα ποτά μας και κατά αυτόν τον τρόπο είχαμε και ένα πολύ θετικό αντίκτυπο και σε άλλες αγορές, σε άλλες εξαγωγές μας αλλά λάβουμε υπόψη μα ότι στα πλαίσια των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών πολύ συχνά πρέπει και εμεί να κάνουμε κάποιε εκχωρήσει όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε πολύ καλύτερη προστασία των γεωγραφικών μα ενδείξεων στι ξένε αγορέ, στι οποίε πηγαίνουν τα προϊόντα αυτά, προκειμένου να καταλήγουμε τελικά σε θετικέ για μα συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών. Θα ήθελα τώρα να σα εξηγήσω λίγο περισσότερο για ποιο λόγο οι γεωγραφικέ ενδείξει είναι πάρα πολύ σημαντικέ για τη γεωργία, την οικονομία μα, το εμπόριο και γενικότερα την απασχόληση. Ας μην ξεχνάμε ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν ανήκουν πλέον μόνο σε δύο-τρία κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τότε υπάρχει να χρησιμοποιεί ένα γενικότερο πανευρωπαϊκό καθεστώ από τη δεκαετία του 90 υπάρχουν όλο και περισσότερε χώρε οι οποίε θέλουν να συμμετέχουν στο σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων. Κάθε κράτο μέλο πλέον τη Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει ένα τουλάχιστον προϊόν γεωγραφική ένδειξη. Δεν αφαιρόμαστε λοιπόν πλέον μόνο στι σαμπάνιε, στο σκοτσέζικο ουίσκι ή στο προσούτο τη Πάρμα, αλλά έχουμε και πάρα πολλά προϊόντα από τη Μάλτα, τη Δανία, την Λετωνία, από πάρα πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλε τι χώρε, όπω σα είπα, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συνολικά έχουμε καταλήξει σε 3.018 γεωγραφικέ ενδείξει. Υπάρχει μια πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία όσον αφορά αυτέ τι γεωγραφικέ ενδείξει. Αν θέλετε, δεν είμαστε πάρα πολύ δυνατοί εμεί σε κάποια πολύ βασικά προϊόντα ω Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά περισσότερο στην παραγωγή κάποιων πολύ ποιοτικών προϊόντων, τα οποία χαίρουν ιδιαίτερη υψηλή φήμη σε ξένε αγορέ. Αναφερθήκατε επίσης και στον Υπουργό Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είχε έρθει στην Επιτροπή σας το Δεκέμβριο. Και ξέρετε ότι είναι έτοιμοι οι ξένοι εταίροι μας να καταβάλουν ένα πολύ σημαντικό αντίτιμο προκειμένου να αγοράσουν τα προϊόντα αυτά και πολλές φορές είδαμε ότι ξεπερνάμε πολλές φορές και δύο φορές την τιμή ενός συμβατικού προϊόντος. Οι γεωγραφικέ ενδείξει ανταστοιχούν λοιπόν σε προϊόντα τα οποία παράγονται από μικρού συνεταιρισμού από μικρού γεωργού και επίση αντιστοιχούν σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό θέσεων απασχόληση στην Ήπεθρο. Για παράδειγμα το κονσόρσιουμ για το Παρμιτζάνο Ρετζάνο απασχολεί πάνω από 50.000 ανθρώπου. Ο συνεταιρισμό ε, για την παραγωγή του τυριού κοντέ στη Γαλλία περίπου 10.000 άτομα και το καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάρα πολλέ θέσει απασχόληση εξαρτώνται στην Ήπεθρο από την παραγωγή προϊόντων που καλύπτονται από γεωγραφικέ ενδείξει. Σε στο συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθο, κλείνει συνεχώ το μικρόφωνο μου. Ενδεχομένω οι συναδελφοί μου από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να θέλουν να, σταμα... να με κάνουν να σταματήσουν να μιλάω. Α δούμε τώρα τι διαπραγματευόμαστε. Καλύτερα, καλύτερη προστασία, καλύτερη επιβολή των ε, γεωγραφικών αυτών ενδείξεων, όπως κάνουμε γενικότερα και με τα πνευματικά δικαιώματα. Ξέρετε ότι προβλέπονται εδώ πέρα συγκεκριμένα συστήματα κυρώσεων ή συστήματα παραβιάσεων κάθε φορά που εμφανίζεται κάτι τέτοιο σε ξένους εταίρους. Βλέπετε εδώ πέρα μια, ένα τυρί φέτα το οποίο έχει παρασκευαστεί στην Αυστραλία και ουσιαστικά παρουσιάζεται ως ελληνική φέτα. Έχουμε ένα προσούτο εδώ πέρα στη φωτογραφία το οποίο παρουσιάζεται ως ιταλικό προσούτο. Έχουμε το όνομα μιας εταιρείας με μια ιταλική μάλιστα σημαία και έχουμε εδώ πέρα και δαμάσκηνα από την Αζό που κανονικά θα προέρχονταν από την περιοχή Αγκουλέμ κοντά στο Κονιάκ αλλά αυτά είναι δαμάσκηνα που πολλούνται τελικά στην Ιαπωνία και παράγονται στην Καλιφόρνια. Εδώ πέρα ουσιαστικά έχουμε μια κατάχρηση των γεωγραφικών αυτών ενδείξεων που οδηγεί σε παραπλάνηση του καταναλωτή και οδηγεί σε πολύ σημαντική οικονομική ζημία για τους παραγωγούς μας. Να σας δώσω ακόμα κάποια παραδείγματα. Βλέπετε εδώ πέρα κάποια προϊόντα τα οποία παραπέμπουν σε ευρωπαϊκά ονόματα. Για παράδειγμα βλέπετε εδώ πέρα Μπορντό, κατά λέξη βαριεστημένη ελαφίνα, το οποίο παραπέμπει βέβαια στο τοπονίμιο Μπορντό, η Γκότροτή. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι προσπαθούν πάλι να χρησιμοποιήσουν κάποια πολύ φημισμένα ευρωπαϊκά ονόματα βάλουν κατά της καλής φήμης των ε, προϊόντων αυτών βέβαια γιατί πολύ συχνά τα προϊόντα τα οποία πολλούνται έτσι, τα παραποιημένα αυτά προϊόντα είναι πολύ χαμηλής ποιότητας ή τουλάχιστον κατώτερης ποιότητα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Τι προσπαθούμε τώρα εμείς να πετύχουμε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Τέσσερα πράγματα. Ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για τις ονομασίε και τις αγορές μας, Ακολουθούμε εδώ πέρα το άρθρο 32 του ΠΟΕ. Έχουμε τη συμφωνία TRIPS, την οποία χρησιμοποιούμε. Έχουμε μια τη βολή επίσης ε, των γεωγραφικών ε, ενδείξεων. Και αυτό το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά είναι ότι αν χρειάζεται Ευρωπαϊκή Παραγωγή να πάνε σε Αμερικανικά δικαστήρια για να υποστηρίξουν μια γραφική ένδειξη, αυτό μπορεί να στοιχήσει δεκάδες χιλιάδες ε, ευρώ και πολλοί παραγωγοί μας, όπως σας είπα, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να κάνουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο προβλέπεται αυτή η αυτεπάγγελτη επιβολή των υγραφικών ενδείξεων. Επίσης θέλουμε τα εμπορικά σήματα να μπορούν να συνεπάρχουν μαζί με τις γεωγραφικές ενδείξεις και αυτό προσπαθούμε να το περάσουμε στα πλαίσια των Συμφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών σύμφωνα με, την, με τον κανονισμό TRIPS του ΠΟΕ. Θέλουμε επίσης να έχουμε μία προστασία μεμονωμένων γεωγραφικών ενδείξεων μέσω διμερών συμφωνιών. Όσον αφορά τώρα τις πολυμερείς μας συμφωνίες, προσπαθούμε να πετύχουμε καλύτερες συμφωνίες στα πλαίσια του ΠΟΕ. Αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση στα πλαίσια της αναπτυξιακής ατζέντα της ΔΟΧΑ. Δεν έχει σημειωθεί όμως αρκετή πρόοδος και ούτε πρόοδο είχαμε τελικά και στην Υπουργική Διάσκεψη του Ναϊρόμπι. Παρ' όλα αυτά όμως Κάτι θετικό το οποίο έχουμε είναι η Σύμβαση της Λισαβόνας στα πλαίσια του WIPO, του Διεθνούς Οργανισμού Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, μια πολυμερής ουσιαστικά συμφωνία, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν τα κράτη-μέλη και να προστατεύουν τις γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν ενταχθεί σε αυτή τη συμφωνία. Έχουμε επίσης σε διμερές επίπεδο πάρα πολλές συμφωνίες για την προστασία συγκεκριμένων προϊόντων, όπως για παράδειγμα κρασί ή αλκοολούχα ποτά, με χώρες όπως η Αυστραλία ή οι Ηνωμένε Πολιτείες. Επίσης, Βλέπετε εδώ πέρα αρκετέ χώρε με τι οποίε διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή ευρύτερε συμφωνίε προστασία γεωγραφικών ενδείξεων στα πλαίσια κυρίω συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Καναδά, Κολομβία, Περού είναι κάποια παραδείγματα, αλλά και με την Ελβετία, το Μαρόκο και την Ουκρανία διαπραγματευόμαστε. Και έχουμε επίση και γεωγραφικέ ενδείξει στα πλαίσια των εξελίξεων διαπραγματεύσεων των εμπορικών που κάνουμε με χώρε όπω το Βιετνάμ, Ολοκληρώθηκε πρόσφατα αυτή η συμφωνία και καταφέρνουμε να προστατεύσουμε περίπου 150 Ευρωπαϊκέ γεωγραφικέ ενδείξει. Έχουμε επίση και την Ιαπωνία, μια πολύ σημαντική αγορά για τι γεωγραφικέ μα ενδείξει. Ινδία, Μερκοσούρ, Νορβηγία και βέβαια και οι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου στα πλαίσια του TTIP προσπαθούμε πάλι να προστατεύσουμε τι περισσότερε γεωγραφικέ μα ενδείξει. Και στο μέλλον θα έχουμε την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία, το Μεξικό, τη Χίλη θα είναι πολύ σημαντικές οι γεωγραφικές προελεύσεις για όλες αυτές τις χώρες. Και κλείνοντας, Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια για την TTIP, όπου οι ονομασίες γεωγραφικής προέλευσης φαίνεται να λαμβάνουν μια μεγάλη σημασία και να γίνονται μήλων της έρευνας στη διαπραγμάτευση. Εμείς επιδιώκουμε στη TTIP ιδιαίτερα υψηλή προστασία για τα τρόφιμα μας, ε, τήρηση από τις ε, κρατικές υπηρεσίες των ονομασιών προελεύσεων, χρειάζεται να καταφεύγουμε στα Αμερικανικά δικαστήρια και άλλων συμβόλων βεβαίω ε, προστασία, ονομάτων, σημεών κτλ. Και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν με σύγκρουση επωνυμιών με γνωστές αμερικανικές επωνυμίες και σήματα. προσπαθήσουμε δε. Ε, ονομασίες προέλευσης που έχουν μείνει και χρησιμοποιούνται στην Αμερικανική αγορά εδώ και χρόνια, όπως τη σαμπάνια, το τοκέ, το πόρτο και το καθεξής, να τα οφήσουμε σταδιακά προς την κατάργηση. Δεν το έχουν δεχθεί ε, στις γενικές διαπραγματεύσεις Αμερικανίου, οπότε θέλουμε να το βάλουμε διμερώς στην TTIP. Είναι κάτι μας απασχολεί εδώ και πολύ και θέλω εταίρως να υπογραμμίσω γιατί πολλή προπαγάνδα ακούγεται στα μέσα για την TIP και τις ονομασίες προέλευση, ότι δεν ζητούμε αλλαγές σημαντικές στο αμερικανικό σύστημα, ούτε θέλουμε να επιβάλλουμε το δικό μας σύστημα των ονομασιών προέλευσης που είναι όπως και να το κάνουμε ιδιάζουν ούτε να επιβάλλουμε δικούς μας, δικές μας ονομασίες ή να προστατεύσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ονόματα που δεν προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καμαμπέρ, μπρι, ε, τσορίσο, μοτσαρέλα, προβολόνε, ό,τι και να σας λέει η αντίθετη προπαγάνδα, δεν προσπαθούμε να προστατεύσουμε αυτά. Μια από τις ηρωνίες, δε, τραϊκή ηρωνία της TTIP, είναι ότι παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιταχθεί κατά τρόπο απερίφραστο στην προστασία των γεωγραφικών προελεύσεων ε, έχουν διμερεί συμφωνίες με ονομασίες προελεύσεως που δεν λέγονται ονομασίες προελεύσεως αλλά ε, προστατευόμενες ονομασίες όπως είναι το whisky του Tennessee Φερρυπίν και στις άλλες διμερείς συμφωνίες ε, τις έχουν εισαγάγει. Εν πάση όλα αυτά θα περάσουν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα προϊόντα, το προϊόν αυτής της διαπραγματεύσεως θέλουμε να έχουμε ένα περιθώριο για υποχωρήσει το χρήστη να κάνουμε για άλλα γεωργικά προϊόντα. Οι Αμερικανοί πάντως προς το παρόν αντιδρούν, δεν θέλουν να διαπραγματευθούν ε, γεωγραφικές ενδείξεις και μάλιστα ζητούν και το περιορισμό, τη μείωση του δικού μας επίπεδου προστασίας για τα δικά τους προϊόντα, κάτι το οποίο αποκλείεται να δεχθούμε. Άρα έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μα. Αλλά θέλουμε ένα καλό αποτέλεσμα για τι γεωγραφικέ ενδείξεις, ώστε να είναι η συμφωνία τη στο δυνατόν πιο ισορροπημένη και καλή. Και καθώ προχωρούμε τώρα κάπου στο ε, μέσον, όπως λέμε, τη παιδιά για το διαπραγματεύσει, έχουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτέ. Και η Επιτροπή σα πιστεύω, θα συνεχίσει να μας υποστηρίζει να μας υποστηρίζει σε ένα φιλόδοξο εγχείρημα σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις στην TTIP αλλά και σε άλλες συμφωνίες. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα πρόεδρε και βεβαίως είμαι στη θέση των βουλευτών για να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση. Δεν υπερεύει το χρόνο σας. Ούτε πρόκειται να σας απενεργοποιήσω το μικρόφωνο. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος κάνει κάτι τέτοιο. Έχουμε 7 ή 8 ομιλητές που δήλωσαν ενδιαφέρον. Κανείς άλλος. 1,5 λεπτό παρακαλώ το πολύ για να προλάβει και ο Γενικός Διευθυντής να απαντήσει. Αλλά πιστά παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο σας. Κύριε Σλάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την ευχαριστήσω για τις εξηγήσεις. Σε ό,τι αφορά το TTIP, Ε, ξέρετε ότι αν δεν βρούμε λύσεις και αν δεν εισακουστούν τα αιτήματά μας θα καταψηφίσουμε. Τώρα, για τις γεωγραφικές ενδείξεις ε, και κυρίως ε, για το ζαμπό της Πάρμας. Σας είχα στείλει και προφορική ερώτηση. Έχουμε πολλές απάτες εδώ. Πρόκειται για ζαμπόν που παράγεται από χείρους που δεν έχουν καν ε, εκτραφεί στην ε, Ιταλία, στην Πάρμα, αλλά στις κάτω χώρες. Και παρόλα αυτά φέρνουν την ονομασία Ζαμπόν Πάρμας. Υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου και επιθεώρησης, γιατί απάτες αντίστοιχε με αυτές που γίνονται με το ζαμπόν και τα γουρούνια μπορούν να συμβούν για άλλα προϊόντα και τελικά ποιος πληρώνει ο καταναλωτής. Παρακαλώ, θα είμαι πολύ αυστηρός. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριος Δες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόλις μου έδωσε ένα άρθρο, μια... μου έστειλε μάλλον ένα άρθρο μια συνεργάτης για νέα ρεκόρ εξαγωγών 8,9 δισεκατομμυρίων ευρώ βαβαρικών γεωργικών προϊόντων στα λοιπά ευρωπαϊκά κράτη αλλά και πέραν αυτών. Εξαγωγές λοιπόν, μεγάλο κομμάτι των οποίων μπόρεσαν να απολυθούν ακριβώς επειδή έχουν καλό ε, καλή γεωγραφική ένδειξη προελεύσεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Είναι σημαντικό και για την TIP και ένα συνάδελφος από τον Bundestag μου είπε όταν είδαμε αυτές τις ε, παραποίησεις ότι πρέπει να φροντίζουμε να βάζουμε και την εθνική σημαία πάνω σε τέτοια προϊόντα γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολο να αναγνωρίζεται η παραποίηση. Βέβαια το βρετανικό η Βρετανική Αυτοκρατορία είχε ζητήσει παλαιότερα να μπαίνει η γερμανική σημαία πάνω στα γερμανικά προϊόντα για να εμποδίσει την κυκλοφορία τους. Πιστεύω ότι αυτό πια δεν ισχύει. Η κυρία Ράς Γκαρσία. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και το Γενικό Διευθυντή για τις εξηγήσεις. Έχω δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτον, η συμφωνία του 2006 με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, άφησε για 17 ονομασίες προέλευσης με τη Μάλαγα, το Χερές, το Πόρτο και άλλα πολλά προϊόντα μέσα με, να, μην τηρούνται και να μην γίνονται σεβαστά. Θα απαιτήσετε την εφαρμογή αυτών των γεωργικών ενδείξεων στην Νέα Συμφωνία και είναι κόκκινη γραμμή συμφωνία για τις γεωγραφικές ενδείξεις προκειμένου να δεχτούμε ένα γενικότερο γεωργικό πακέτο στο TTIP. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις και παρακαλώ περιμένω απάντηση. Λαμπρά, κύριε Ράσγκαρσία, τηρήστε το χρόνο σας. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σύντομες ερωτήσει. Με την πρώτη θα υποστηρίξω τόσο επί κυρία Πύρη. Για την ε, καθαρότητα της γεωγραφικής ένδειξης όπου ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί μας λένε καλά μην ε, ε, ενοχλείστε πάρα πολύ, μπορεί να το λέμε ε, ζαμπόν τυρόλου, αλλά το χοιρινό από το οποίο γίνεται το ζαμπόν αυτό δεν έχει εκτραφεί στο τυρόλο. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο ίσως θα ήταν καλό να κάνουμε μια ε, έφοδο, μια εφόρμηση διαφάνειας θα έλεγα, για να κάνουν αυτή τη διαφεροποίηση μεταξύ του Made in Europe και του Made in United States. Έχετε εσείς κάποιες τις προτάσεις, έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μας ε, να στηρίξουμε την Ευρώπη ως χώρο παραγωγής και πού θα βρεθεί η ισορροπία και η λύση εκείνη η οποία θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ. Κύριε Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω με τι ταχύτητα διεκπεραιώνεται τις αιτήσει, γιατί 18 αιτήσει στάλθηκαν από την Κροατία που είναι νέα χώρα μέλος. Μέχρι στιγμής 7 έχουν γίνει δεκτές. Μερικές απαιτήσει ίσως είναι προβληματικές ε, γιατί και μάλιστα θα πρέπει να συμπληρωθούν. Ε, επίσης, τι γίνεται με την ονομασία προέλευσης και τη γεωγραφική έδειξη και η σχέση μεταξύ των δύο. Είναι σημαντικό το λάχανο από το Βαρασδίν να φέρει και το όνομα της πόλης στην οποία παράγεται. Και αυτή η πόλη, το Βαρασδίν, βρίσκεται στην Κροατία. Και ε, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να φαίνεται ότι αυτό το λάχανο από το Βαρασδίν είναι ε, προέλευση Κροατίας. Πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα. Ο κύριος Αντρία, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσυπογράψω την ερώτηση της κυρίας Σεράς Καρσία. 17 ονομασίες έμειναν χωρίς λύση στην προηγούμενη συμφωνία για ημιγενώσιμα. Επίσης, ευχαριστώ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Μας είπατε όμως ότι οι Αμερικανοί δεν θέλουν νέες διαπραγματεύσεις για τις γεωγραφικές ενδείξεις, άρα θα δημιουργηθεί πρόβλημα, θα δημιουργηθεί αδιέξοδο και στην συμφωνία ε, του, του TTIP υπάρχει κάποια πρόοδος, γιατί θα ήταν παράδοξο δεδομένης άνησής τους να συμπεριλάβουν τις γεωργικές ενδείξεις μέσα. Μήπως ε, ε, ακριβώς χρησιμοποιούν συγκεκριμένη διαπραγματευτική στρατηγική γνωρίζοντας ότι θα προσκρούσουμε στις γεωγραφικές ενδείξεις και τις κρατάνε αυτά, τις κρατούν για το τέλος προκειμένου να μας κάνουν να δεχτούμε άλλες παραχωρήσεις σε άλλα θέματα. Ε, θα πρέπει όμως να ξεπεράσουμε το διέξοδο ε, των γεωγραφικών ενδείξεων στις διαπραγματεύσεις. Ε, τι σημαίνει αυτό, ότι αν παραμείνει το διέξοδο θα σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις και στα υπόλοιπα θέματα. Ο κύριος Άγνιου. Η Επιτροπή βαδίζει μέσα σε ένα ναρκοπέδιο, αμφίβολα. Αναφερθήκατε στο Τσένταρ. Ωραία. Το Τσέσιρ που είναι επίση μια επαρχία με πάρα πολλέ αγελάδε και μπορεί να θελήσουν και αυτοί να πάρουν γεωγραφική ένδειξη. Και μετά πάμε σε περιοχές όπως το Τζόρισι που έχει ποικιλίε ζώων, ράτσα αγελάδα και πολλά άλλα μπορώ να σας αναφέρω ως προϊόντα τοπικά. Το Yorkshire Pudding όπως και πολλά άλλα επί που είναι όμως συνταγές και οι μόνοι που μπορούν να τα λύσουν αυτά ως προβλήματα είναι ε, τα κράτη-μέλη. Με κανένα άλλο τρόπο δεν μπορείτε να βρείτε λύση. Φλάναγκαν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αναφερθήκατε σε φήμες σχετικές με την TTIP. Γιατί λέτε φήμες, μήπως επειδή υπήρξε κενό ενημέρωσης και εν κενό ενημερώσεως προκύπτουν φήμες. Μήπως θα ήταν σκόπιμο εσείς να μας ενημερώνετε πιο τακτικά και να μας δώσετε στοιχεία για τις εξαγωγές του κυρίου Ντέσα από την <laughs> Βαβαρία θα ήθελα να πω ότι η δική μου περιοχή φτιάχνει καταπληκτική μπύρα και μπράβο τους. Κυρία Αγγιλέρα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και το Γενικό Διευθυντή για τις εξηγήσει. Και εγώ έχω συγκεκριμένη ερώτηση. Η ιστορία των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρώπης ήταν μια success story. Και μάλιστα στην Ολομέλεια εγκρίναμε έκθεση πρωτοβουλίας, ώστε το μοντέλο μας για τις γεωγραφικές ενδείξεις να το μεταφέρουμε και σε παραγωγές που δεν αφορούν τρόφιμα. Υπάρχει κάποια πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη μετάθεση αυτού του μοντέλου και σε άλλα προϊόντα εκτό των τροφίμων. Τώρα, μία συγκεκριμένη ερώτηση. Είπατε ότι επιχειρήσατε κάλυψη των κυβερνητικών ενδείξεων από προστασία στι διαπραγματεύσει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και είπατε ότι δεν ε, διαπιστώσατε καμία πρόοδο. Γιατί εκεί ήταν το κατάλληλο φόρουμ για να επιδιωχθεί προστασία, αλλά από ό,τι κατάλαβα από τι εξηγήσει ε, δεν εξασφαλίστηκε η προστασία αυτή στον ΠΟΕ. Η κυρία Εράς και ο κύριος Άντριου σας έθεσαν μια ερώτηση για το TTIP. Οι γεωγραφικές ενδείξεις θα είναι κόκκινη γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Διαπραγματεύσης του TTIP. Δεν κατάλαβα από τις εξηγήσεις που μας δώσετε πριν αν όντως είναι κόκκινη γραμμή οι γεωγραφικές ενδείξεις της διαπραγματεύσης. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κλάρκ για την συνοπτική αλλά μεστή παρουσίαση που μας βοήθησε να εξοικειωθούμε κάπως με το πρόβλημα. Πήγα πρόσφατα στι Ηνωμένε Πολιτείε, ενδιαφέρουσα επίσκεψη και θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορούμε, μπορεί να σταθεί το επιχείρημά μας στο γεωγραφικό αναδείξεων απέναντι στο δικό τους επιχείρημα. Γιατί όταν εμεί μιλούμε για γεωγραφικέ ενδείξει, εκείνε μα προτάσουν το επιχείρημα του εμπορικού σήματο. Είναι αρκετά α, σημαντικό επιχείρημα. Είναι συμβατά μεταξύ του δύο. Θα μπορούσαν να συνεπάρχουν τα εμπορικά σήματα με τι γεωγραφικέ ενδείξει. Και επειδή εγώ κατάγομαι από μια περιοχή που μόλι μπήκαμε σε αυτή, αυτό το χώρο των ονομασιών προέλευση και των προστατευμένων ενδείξεων, μας αρέσει αυτό το θέμα, αλλά δεν δεν ξέρω αν θα θέλαμε όλα τα προϊόντα και όλοι οι τομεί να γίνουν ε, εχμάλωτοι στι διαπραγματεύσει και το διεξόδου που θα δημιουργηθεί ενδεχομένω από τι γεωγραφικέ ενδείξει. Ευχαριστώ κύριο Τσούλο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Όσον αφορά την συμφωνία TTIP, αν καταφέρναμε να προστατεύσουμε τις γεωγραφικές ενδείξεις ξέρετε ότι υπάρχουν 3.000 ε, τέτοιες προστατευόμενες ονομασίε, πώς θα προστατευόντουσαν όμω, ποια κριτήρια θα χρησιμοποιούσαν προκειμένου να επιλέξουμε κάποιες ενδείξεις, να προστατεύσουμε κάποιες ενδείξεις και κάποιες άλλε όχι. Ευχαριστώ. Και εγώ μία σύντομη ερώτηση. Μήπως το παρατραβάμε με τις γεωργικές ενδείξεις. Ξέρω ότι αγαπάμε τα προϊόντα μα. αλλά το καλύτερο σημάδι, η καλύτερη εγγύηση είναι η ποιότητα. Δεν θα πρέπει σε αυτό να επικεντρωθούμε. Στη γεύση, στην ποιότητα. Μήπως αν μείνουμε τόσο στις γεωγραφικές ενδείξεις θα περιορίσουμε έτσι αναγκαστικά τις εξαγωγές μας. Δεν ξέρω, μπορεί να αγγίζω εδώ ευαίσθητες χορδές και πράγματα που πονάνε. Και σίγουρα στο θέμα του TTIP θα επανέλθουμε γιατί σίγουρα είναι λυπείς οι πληροφορίες που έχουμε λάβει και θα πρέπει να συμπληρωθούν αυτές όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από αυτή σίγουρα. Thank you. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το φόρκα το πολωνικό είναι από τα πιο γνωστά. Α, η βότκα η πολωνική, συγγνώμη, είναι από τις πιο γνωστές ε, ε, ονομασίες ε, από τις πιο γνωστές γεωγραφικές ενδείξεις αν θέλετε να ξέρετε. Έχει πάρα πολύ καλές πωλήσει. Ας προσπαθήσω να απαντήσω όμω στις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις ώστε να τον περισσότερες. Πολλοί από εσά ε, συμφωνείτε ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις έχουν κέρια σημασία για τις διαπραγματεύσεις μας, όντως καθώς εκπροσωπούν πολύ σημαντικό ε, ποσοστό των εξαγωγών και του εξαγωγικού δυναμικού των προϊόντων μας αποτελούν μια επιτυχία της ε, προσπάθειας εξαγωγικής των γεωργικών ε, προϊόντων. Και αυτό όσο το δυνατό, και γι' αυτό όσο δυνατόν περισσότερα προϊόντα, τρόφιμα, ποτά κτλ. μπορούμε να εξαγάγουμε στην ε, Γεωργία, στην, στις ΗΠΑ, στην την Ιαπωνία, την Κίνα, τόσο το καλύτερο. Τώρα για το ζαμό της Πάρμας που ρωτήσατε νωρίτερα, που μπορεί να προέρχεται από ε, κρέας χείρων που δεν έχουν εκτραφεί στην Πάρμα. Όχι, δεν επιτρέπεται αυτό. Πρέπει να έχει γίνει εκτροφή σε ένα συγκεκριμένο χώρο και μια συγκεκριμένη διαμόρφωση γεωγραφική ιταλικών περιοχών. Παρά τις όποιες φήμες λοιπόν δεν είναι δυνατόν να είναι εισαγόμενα από άλλες περιοχές του κόσμου τα ζώα και μετά να τα βαφτίζει η Ιταλία ε, Ζαμπον Πάρμας. Πολλοί από σας αναφέρθηκαν ε, στα ημιγενώσιμα ονόματα Ίνους, Πολιτείς, κυρία Ράντσα Γκαρσία, αν δεν την εκείνη, η οποία μας είπε ότι υπάρχει, υπάρχει τέτοιο θέμα, έχουμε μια πρώτη συμφωνία θα προχωρήσουμε σε μια σταδιακή απαγόρευση των 17 αυτά ονομασιών. Δεν έχουν ακόμα αποδεχθεί τα πάντα οι Αμερικανοί. Δεν έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο πίεση σε μια διμερή συμφωνία να επιβάλλουμε ε, τη λύση που θέλουμε. Μόνο χάρη στη DTIP μπορούμε να πιέσουμε για τα 17 αυτά, για τα 17, αυτές ονομασίες. Για τον κύριο Γιάρς. που μας αν μπορούμε να έχουμε γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προελεύσεως. Δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες. Οι κανόνες προελεύσεως ισχύουν για κάθε ε, προϊόν, για, τα, για τις επωνυμίες δεν έχουμε πρόβλημα τη σχέση με την προέλευση με τους Αμερικανούς. Οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι μια διαφορετική μονάδα μέτρηση έχει να κάνει με την βιομηχανική ιδιοκτησία. Η γεωγραφική ένδειξη βεβαίως και κάθε ευρωπαϊκό προϊόν θα καταγράφει ότι προέρχεται από την Ευρώπη ή από ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η γεωγραφική ένδειξη δηλαδή είναι ως προς τη σύλληψη της διαφορετική ένδειξη. Άλλη ερώτηση. Τον αντιπρόεδρο να μην τον απατώμε για το αν μπορεί να αποτελέσουν κόκκινη γραμμή για τις διαπραγματεύσεις TTIP, γεωγραφικές ενδείξεις, για, τις, για τα γεωργικά προϊόντα ενδεχομένω ως προϋπόθεση, δηλαδή για την ολοκλήρωση του πακέτου σχετικού με τη γεωργία ή εν όλο. Δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή, είναι πρόημο. Πάντως εντολή του Συμβουλίου καθιστά απόλυτα σαφές ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις πρέπει να είναι μέρος της TTIP. Τα δε μηνύματα που ακούω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παγίως μου λένε ότι δεν είναι νοητή μια τέτοια επιχωρήση της γεωγραφικής ένδειξης. Στις γεωγραφικές διαπραγματεύσεις πάντως για μένα θα ήταν αδιανόητο να καταλήξω σε θέματα γεωγραφικά, συμφωνία, σε συμφωνία χωρίς γεωγραφικές ενδείξεις. Γιατί αυτό είναι, αν θέλετε, το κύριο, μαζί με τα γαλακτοκομικά, επιθετικό συμφέρον της Ευρώπης σε μια TTIP και δει στη γεωργική της, στο γεωργικό της σκέλος, αλλά και σε ολόκληρη τη συμφωνία. Για τον κύριο Νίκολσον. Ελπίζω να μην τον έπεισαν ε, ή να μην τον γίτεσαν οι Αμερικανοί όταν επισκέφθηκε τη χώρα τους. Έχουν ένα ταλέντο να πείθουν ότι το σύστημα των, ε, του trademark, δηλαδή της προστατευόμενης επωνυμίας, αρκεί. Δεν αρκεί γιατί δεν επιτρέπει επιτρέπει υψηλό βαθμό προστασίας για τα τρόφιμα. Το σύστημα των ονομασιών, των επωνυμιών, έχει χαμηλό επίπεδο προστασίας ως εμπορική επωνυμία για τις γεωγραφικές ενδείξεις και γι' αυτό δεν καλύπτουμε μέσα από το σύστημα των επωνυμιών τη γεωγραφική ένδειξη και ε, δεν μπορούμε να την προστατέψουμε αν δεν καταφύγουμε σε αμερικανικά δικαστήρια, πράγμα το οποίο σημαίνει τεράστιο κόστος για την επίλυση τέτοιων διαφορών. Άρα δεν μας καλύπτουν ε, ούτε σε επίπεδο προστασίας, ούτε και σε επίπεδο ε, σεβασμού ε, τα ε, οι επωνυμίες αμερικανικές, το σύστημα των επωνυμιών σε σχέση με τις γεωγραφικές ενδείξεις για τον κύριο Άγνιου που μας είπε ότι έχουμε πατήσει στην αρκοπέδιο. Είναι πολύ ευαίσθητος τομέας γεωγραφικής ενδείξης, το δέχομαι. Είναι θέμα παράδοσης, είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα το τι τρώμε ξεπερνά σε μεγάλο βαθμό τη σημασία της ε, πνευματικής διοκτησίας. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά οι γεωγραφικές ενδείξεις στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί, έχουν καταχωρηθεί, καταχωριστεί, έχουν αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο. Η γεωγραφική ένδειξη πρώτα αναγνωρίζεται ή το τσένταρι παραδείγματι, για να μιλήσουμε για το σκοτσέζικο ουίσκι, ναι, το Yorkshire Pudding δεν είναι γεωγραφική ένδειξη, αν και εγώ δεν έχω καταλήξει ότι θα έπρεπε να είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρώτα αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται σε εθνικό επίπεδο και μετά το κράτος μέλος αποστέλει τη γεωγραφική ένδειξη για πανευρωπαϊκή προστασία. Και έτσι όχι μόνο στον Εμένο Βασίλειο ή ε, την Αυστρία, αλλά για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία εάν θέλουμε να προωθούμε και να πολλούμε τα προϊόντα μας σωστά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στο ένα κράτος μέλος από το οποίο προέρχονται. Για το αν είναι ρεαλιστικό να επιδιώκεται προστασία σε συμφωνίες με τρίτες χώρες των 7.000 και γεωγραφικών ενδείξεων, η απάντηση είναι αρνητική. Στις περισσότερες εμπορικές συμφωνίες προσπαθούμε να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο κατάλογο 150-200 το πολύ σημαντικών εμπορικά γεωγραφικών ενδείξεων η μέγιστη πλειονότητα των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βγαίνει καν από το κράτος μέλος το οποίο έχει γεννηθεί η γεωγραφική ένδειξη και έχει ε, αναγνωριστεί. 150 ε, με 200 μπορεί να έχουν σημασία εμπορική μόνο και γι' αυτό έχουμε έναν ε, κατάλογο. Βέβαια, σε σχέση με τις όμορες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρας όπως είναι η Ελβετία, συνάπτουμε συμφωνίες που καλύπτουν ένα πολύ ευρύτερο κατάλογο, γιατί δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων χωρίς καλή συνεργασία με τους εταίρους μας. Επίσης ο κύριος Φλάνναγκαν ε, που έκανε το σχόλιο για την TTIP και τα σχόλια. Σε λίγο θα πρέπει να ολοκληρώνετε λέει ο γραμματέας. Ναι, Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει μια στρατηγική προσπαθεί να υποβαθμίσει τη σημασία των γεωγραφικών ενδείξεων και λέει ότι δεν αρκούν για την ζήτηση, ότι δεν υπάρχει πραγματικό εμπορικό συμφέρον ως προς την διατήρηση των γεωγραφικών ενδείξεων. Υπάρχουν πολλοί κυρίως στυροκόμοι γαλακτοκομικός τομέας που χρόνια τώρα παράγουν εντό εισαγωγικών φέτα ή γκοργοντζόλα ή άλλα τυριά και δεν θέλουν να βγουν από αυτή την κατάσταση που τους επιτρέπει την ασυνοσία. Κάποιοι που μπορεί να βάζουν και η Ιταλική σημαία στο τυρί τους ακόμα, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Εκμεταλλεύονται τη φήμη σημαντικών Ιταλικών ε, τυριών της Ευρώπης. Και σταματώ εδώ, Πρόεδρε, γιατί η Γερμανία τελείωσε. Σας ευχαριστούμε κύριε Γενική Διευθυντά. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση που μας κάνατε και δεν είναι η πρώτη φορά. Μας έχετε συνηθίσει σε ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Σίγουρα ε, ο Σονούπο θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά. Και οι δυσκολίε θα αρχίσουν από τη στιγμή που καταλήξουμε σε αυτό το σύντομο κατάλογο 150 με 300 προϊόντων. Τότε θα αρχίσουν τα δύσκολα, όταν καταλήξουμε στις γεωγραφικές ενδείξεις που θα προστατεύσουμε. Φαντάζομαι μας περιμένουν εκτενέστατες ε, συζητήσεις για το TTIP. Επόμενη συνεδρία 22 και 23 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ. Καταφέραμε και διεκπεράσαμε την ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ και του εκπροσώπους τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό σα βράδυ.